Mes chers collègues, bonjour. On va y aller. Bonjour. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Monsieur Wim van de Kamp, on vous attend. Κύριε Wim van de Kamp, σας περιμένουμε. Κύριε Βάσκη, καλημέρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ελπίζω όλοι σας να περάσατε ευχαριστές διακοπές, να φορτίσατε τις μπαταρίες σας για ένα έργο το οποίο μας περιμένει πολύ πλούσιο μέσα στο επόμενο έτος. Μας περιμένει ένα χρόνος γεμάτος δουλειά. Δεν ξέρω κυρία Φώστερ ε, αν θα είναι πολύ αν δεν έχετε παρατηρήσεις και αντιρρήσει για την ημερησία διάταξη, το σχέδιο ημερησία διάταξη μπορεί να εγκριθεί. Τα πρακτικά της ε, συνεδρίασης 9 και 10 Ιουλίου του 2018 επίσης εγκρίνονται, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, η σχολικές ε, διακοπές χαρακτηρίστηκαν δυστυχώς από ένα τρομακτικό περιστατικό στην Ιταλία 14 Αυγούστου η γέφυρα Μοράντι του αυτοκινητοδρόμου Α10 που συνδέει τη Γιάννοβα με τη Σαβόνα και τη Βεντιμίλια κατέρευσε. Επίσημος απολογισμός ε, της τραγωδίας δυστυχώς είναι 45 νεκροί. Θα ήθελα λοιπόν εκ μέρους όλων μας ε, να απευθύνω τα ειλικρινά μου συλληπιτήρια στη συγγενείς των θυμάτων. Σε αυτόν τον τραγικό απολογισμό ε, προστίθενται εκατοντάδες άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους ε, όταν έπεσε αυτή η γέφυρα στην κατοικημένη περιοχή που βρισκόταν από κάτω. Μια ολόκληρη γειτονιά τώρα έχει ερημωθεί. Αυτό επηρεάζει τις επιχειρήσεις, τα καταστήματα, την καθημερινότητα των ε, αγαπητών μας ε, Ευρωπαίων γειτόνων για αρκετό χρόνο. Θα ήθελα λοιπόν να υπενθυμίσω ότι θα έχουν όλοι μας την αλληλεγγύη και τη στήριξη. Όσον αφορά τον τομέα των χρηματοδοτήσεων, η Επιτροπή μας πάντα ε, μιλούσε με μία ενιαία φωνή ώστε να διασφαλίζει τη χρηματοδότηση ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υποδομές. Υποδομές ε, που πρέπει να είναι ασφαλείς και σύγχρονες. Ιδιαίτερα στον τομέα των διακρατικών ευρωπαϊκών δικτύων. Θα συνεχίσουμε στην ίδια οδό με όλο και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα μετά από αυτή την καταστροφή. Επαναλαμβάνω, είναι απαραίτητο οι συμπολίτε μας στην Ευρώπη έχουν το δικαίωμα, χρειάζονται ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές που να τους βοηθούν να ζουν την καθημερινότητά τους με ασφάλεια. Στο πλαίσιο των εργασιών μας για τους μηχανισμούς χρηματοδότησης για τις υποδομές θα εξετάσουμε με προσοχή τα μέτρα που υλοποιούνται για την ασφάλεια των υποδομών μας. Η έλεγχη, οι υποχρεώσεις, η συντήρηση και η αποσυμφόρηση της οδικής κυκλοφορίας, η φιλοσοφία της πρόληψης και του εξυγχρονισμού των συστημάτων μεταφορών θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεών μας και να ακολουθούνται από πολιτική και δημόσια κρατική δράση. Είναι καθήκον μας. Δεν μπορώ λοιπόν να ξεκινήσω τις εργασίες της Επιτροπής μας χωρίς να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα και για τους συγγενείς τους μετά από αυτό το τραγικό δυστύχημα. Σας καλώ λοιπόν να τηρήσουμε ενός λεπτού Ευχαριστώ. Merci à vous, chers collègues. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Nous allons commencer les votes. Je remercie. Θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Κυρία Ντεμόντε, είδα ότι δεν έχετε κάρτα. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε πρώτα απ' όλα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και όλα τα μέλη της Επιτροπής για την έκφραση αυτή αλληλεγγύης. Ήταν πολύ δύσκολες οι τελευταίες εβδομάδες ε, για τις ζωές που χάθηκαν από ανθρώπους που πήγαιναν διακοπές ή απλά ανθρώπους που πήγαιναν στη δουλειά τους. Είναι πολύ σημαντικό το ότι η Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκφράζει την αλληλεγγύη της και τη δέσμευσή της για το μέλλον να υποστηρίξει την πόλη, της Γένοβας ε, και το μέλλον όλης αυτής της περιοχής ε, που σήμερα βρίσκεται απομονωμένη λόγω αυτής ε, της υποδομής που κατέρευσε θα, δεν έχω την κάρτα μαζί μου οπότε θα ψηφίσω διανάταση χειρό σήμερα ευχαριστώ ευχαριστούμε κυρία Ντεμόντε η γεφύρα της Γένοβας είναι είσοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντική για την πόλη οικονομικά, τουριστικά και από όψη μεταφορών. Εμείς εδώ στην Επιτροπή μας ε, θα αναλάβουμε όλες μας τις ευθύνες, ούτω ώστε να βοηθήσουμε την πόλη αυτή. Γι' αυτό το λόγο θα γίνει μια συζήτηση με τους συντονιστές και εμένα την επόμενη εβδομάδα για το ζήτημα αυτό. Να ευχαριστήσω ξεκινώντας ε, ε, τους διερμηνείς, ε, να τους ευχαριστήσω για τη δουλειά τους. Ξέρω ότι πριν τις διακοπές τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Ελπίζω λοιπόν με την επιστροφή μας ε, στις εργασίες μας να είναι όλα πιο εύκολα και ευχαριστούμε για τη δουλειά σας. Δεν λέμε διερμηνείς, λέμε μεταφραστές. Εσείς αποφασίζετε, λέει η Πρόεδρος. Ξεκινάμε την ψηφοφορία λοιπόν με τον προϋπολογισμό του 2019. Ο κύριος Τέλιτσκα είναι ο εισηγητής και ας κάνουμε μια δοκιμή για να δούμε κατά πόσο έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό, άρχεται ψηφοφορία, τέλος ψηφοφορίας. Υπάρχουν κάποιοι που ήδη ψηφίζουν κατά τόσο νωρίς το πρωί. Λοιπόν, ξεκινάμε. Α, δεν δουλεύει, αλλάξτε θέση. Λειτουργεί. Ελπίζετε, ελπίζω και εγώ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τροπολογία 5382 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5381 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5365 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5366 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53-67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 να το ελέγξουμε την 53-67 άρχεται η ψηφοφορία για την 53-69 λέει η πρόεδρος 67 λάθος 67 πέρας ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Είχατε δίκιο. 53-69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53-70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53-71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53-87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5389 υπέρ κατά 5389 κύριε Βιμ Βαντεκάμπ γυρίστε τη σελίδα ορίστε λοιπόν 5389 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Θέλετε να επαληθεύσουμε την 5389 άρχεται η ψηφοφορία. Καλημέρα κύριε Ερτούγκ. Πέρα της φοβουρία. Απορρίπτεται. Έχετε με εμπιστοσύνη κύριε Βιμ συνεχιζουμε Συνεχίζουμε 53-76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53-73 υπέρ. Κατά. Αποχές. 53,50 53-50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 53-72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 53-51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53-68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53-52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53-53 υπέρ έχει απορριφθεί 53-53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53-86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53-75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53-77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53-85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53-93 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, δεν είναι σαφές. 53-93. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 53-54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53-88 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 5374 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5390 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5364 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5378 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 53-84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53-98 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές να ελέγξουμε την 53-98 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 53-55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53-79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53, 56, 53, 97 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 53, 83 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημες 5357-5396 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 5358 και 5395 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Δύο ταυτόσημες 5359-5394 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 53-91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53-60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53-61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53-62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 53-63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53-80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συνεχίζουμε με τη συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική ε, συγγνώμη, τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τροπολογία 7 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τα μικρή διαφορά. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 33 υπέρ, καμία κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια, κύριε Τέλιτσκα. Εγκρίνεται η έκθεση σας σήμερα το πρωί. Alors, nous continuons. Και συνεχίζουμε λοιπόν. για τη γνωμοδότηση της εμπο για το Ευρώ 5, έγκριση τύπου ε, για τα δίκυκλα, τρίκυκλα και τετράκυκλα. Η συγγήτρια εγώ ίδια. Ξεκινάμε. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε επαλήθευση. Ωραία. Ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ για την τροπολογία 1. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Για τη 2 παρακαλώ. σήκωσε τα χέρια υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, άρα ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Έναρξη ψηφοφορίας για την τροπολογία υπερκμούν 2. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 3, τροπολογία 3, υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Το ΕΛΚ νομίζω τουλάχιστον το λέει, αλλά θα επαληθεύσουμε. Ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίζουμε για την τροπολογία υπαριθμών 3. Πέρας. Και απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 5. Τροπολογία 5. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Θα τις ψηφίσουμε όλες μαζί, θέλετε, unblock. Κάποιοι διαφωνούν, ωστόσο. Λυπάμαι. Από τη 5 μέχρι τη 10 τότε, unblock. Δεν είμαι σίγουρη. Συνεχίζουμε λοιπόν μία-μία ή πέντε παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η έξι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επτά υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οκτώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εννέα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε. Ας επαληθεύσουμε την τροπολογία υπερθμών 11. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Μα αφού σας το είχα πει κύριε Βιμφαντε Κάμπ. Η 12 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Α, συγγνώμη, υπέρ, λέει η πρόεδρος. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται, αλλά άμα θέλετε πολυθεύουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου τώρα, παρακαλώ. Ψηφίζουμε, παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Πέρας. 33 υπέρ. Μία ψήφος κατά. Συμβαίνουν αυτά. Και τρεις αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν η γνωμοδότηση. Και σας ευχαριστώ. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Να συνεχίσουμε λοιπόν με την έκθεση του κυρίου Βιμ Κάμπ. Si vous sortez, s'il vous plaît, sortez. Όποιο θέλει να φύγει, παρακαλώ να φύγει από την αίθουσα και να κάνει ησυχία. Mais il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui a roulé mon truc. Allez, sortez en silence si vous voulez bien. Allez. Monsieur Wim van Κύριε Βίμ van έτοιμος. Αγαπητοί συνάδελφοι. Αν θέλετε να πείτε τα των διακοπών σας με τους συναδέλφους σας, σας παρακαλώ, βγείτε τουλάχιστον έξω από την αίθουσα. Ευχαριστώ. Allez, nous en venons maintenant à και τώρα να περάσουμε λοιπόν στην παρουσίαση μία από τις πιο σημαντικές εκθέσεις μας, μία έκθεση πρωτοβουλία συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Η έκθεση λοιπόν αυτή ε, εξετάζει ένα θέμα για το μέλλον των μεταφορών, την αυτόνομη οδήγηση στις μεταφορές. Έχετε το λόγο, κύριε Σίγητα, κύριε Βιμ Φαντενκάμπ και μετά θα ακούσουμε τους ε, συνεισηγητέ και στη συνέχεια θα ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο, καταρχάς, κυρία Κάμπο. Κυρία Πρόεδρε. Αγαπητή Καριμά. Χαίρομαι που βρισκόμαστε και πάλι λοιπόν όλοι μαζί εδώ. Τα επιστρέψαμε σόι και βλαβή. Η κυρία Γιάλα Σέντερ εγχειρίστηκε, αλλά περπατάει μια χαρά τη βλέπω. Και άρα θεωρώ ότι η διάθεση είναι άριστη. Το είπατε εισαγωγικά λοιπόν κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι όντω πρόκειται για ένα θέμα το οποίο όχι επειδή είμαι εγώ εισηγητής, ε, αλλά επειδή πραγματικά είναι σημαντικό το θέμα αυτό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ παραπάνω πράγματα πέρα από το ελληνικό χρέος, από τα, την φύλαξη των συνόρων. Είναι πολύ παραπάνω και από την πολιτική του ασύλου. Εδώ λοιπόν σήμερα μιλάμε για μια μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη η οποία θα είναι πραγματικά κρίσιμη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο λόγω της ενιαίας αγοράς, αλλά και λόγω της πολιτικής για την καινοτομία και την τεχνολογία. Θα το είδατε και στην έκθεση είναι ότι δεν μιλάω μόνο για τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα, τα γιοταχή, αλλά κυρίως και για τα πλοία, τα τρένα, ακόμα και για την αεροπορία. Γιατί οι εξελίξεις ε, ε, στις και στο, στην τεχνολογία των μετρό είναι τόσο γρήγορη που ήδη είναι πολλά τα τρένα και οι σιδηρόδρομοι που λειτουργούν χωρίς αυτόνομη, χωρίς ε, οδήγηση, χωρίς οδηγό. Είναι τεράστια ο ανταγωνισμό με τη ΣΥΠΑ και με την Κίνα. Μαζί τον Νοέμβριο του 2017 επισκεφτήκαμε το Silicon Valley στη ΣΥΠΑ και εκεί διαπιστώσαμε ότι στο Silicon Valley υπάρχει αίσθηση ότι είναι ηγετική η τεχνολογία αυτή, αλλά θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι τουλάχιστον σε αντίστοιχο επίπεδο και αυτό θα πρέπει πραγματικά να φροντίσουμε να διατηρηθεί. Παράλληλα, διαπιστώνω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αποτινάξει πια αυτό το σύνδρομο κατωτερότητας που έχει, ότι τα ΧΑΙΠΑ πάντα είναι όλοι καλύτεροι και ότι η Κίνα τα κάνει όλα πιο γρήγορα. Αλλά στο θέμα αυτό, και αυτό φαίνεται από την έκθεση CITS του συναδέλφου Βιελή, ότι δεν υπάρχει πραγματικά λόγος να έχουμε αυτό το σύμπλεγμα πλέον. Και βλέπουμε ότι του κυρίως υποστηρίζεται αυτή η τεχνολογική εξέλιξη για να μην κυριαρχήσει πραγματικά αυτό το σύμπλεγμα 28 κρατών μελών. Ε, παράλληλα πρέπει να είμαστε γρήγοροι. Να είμαστε γρήγοροι και αυτό φυσικά η ταχύτητα δεν είναι χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την νομοθεσία, σε ό,τι αφορά το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο είναι απαραίτητο. Πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη ταχύτητα. Να κινηθούμε γρήγορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το βλέπετε ότι και εισαγωγικά έκανα κάποιες παρατηρήσεις στο D της ε, έκθεσης μου. Ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει, κυρία Πρόεδρα. Το θέμα είναι λοιπόν ε, τι θα κάνουμε. Θα το κάνουμε και θα κινηθούμε προς τα εμπρός 28 μαζί ή θα ή, κινηθούμε 28 ξεχωριστά κράτη-μέλη. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παίξει το ρόλο της ε, αποφασιστικά και δυναμικά στο θέμα αυτό. Ελπίζω και στο νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρξει αυτή η αποφασιστικότητα και να σας υπανθυμίσω και την διακήρυξη του Άμστερνταμ του Ιανουαρίου του 2016 στο σημείο ε. Τι αναφέρεται. Ένα σημαντικό σημείο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε είναι η startup, οι νεοφύση αυτές ε, επιχειρήσεις. Ε, υπάρχει και το σχετικό βραβείο, το οποίο και εσείς υποστηρίξατε, αλλά όλη η τεχνολογική ε, καινοτομία σε ό,τι αφορά τα αεροπλάνα, τα γεωτραχή, ε, και όλα τα μέσα μεταφοράς δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε αυτή η ταχύτητα, αυτή η τάση νετορισμό που μας δίνουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Και αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε. Πρόεδρε, να ολοκληρώσω στο σημείο αυτό της εισαγωγική μου παρατηρήσεις. Ξέρετε ότι δεν μπορούν να, ε, να περιληφθούν τα πάντα σε εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας, γιατί έχουμε περιορισμούς ως προς το χώρο, αλλά τις καλές ε, τροπολογίες σίγουρα θα τις ε, υποστηρίξουμε. Να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Κοινωνικών και Οικονομικών Υποθέσεων, η οποία ήδη γνωμοδότησε και θα λάβω υπόψη τα σχόλιά τους. Και με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένω και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων επιτροπών, της ΙΜΚΟ, της Γιούρη, της Ήτρε. Όλες αυτές οι επιτροπές θα γνωμοδοτήσουν. Και ξέρουμε ότι η προστασία δεδομένων, για παράδειγμα, στα αυτοκινούμενα οχήματα, αλλά και η αστική ευθύνη σε περίπτωση αυτοκινούμενων οχημάτων, είναι νομικά ζητήματα, τα οποία προφανώς θα πρέπει να τα εξετάσουμε σε βάθος. Τέλος, Πρόεδρε, ο άνθρωπος πώς θα ζήσει αυτή τη ε, μετάβαση. Στην τελευταία παράγραφο προσπάθησα να βάλω τον ανθρώπινο παράγοντα ως ε, στρεβλωτικό παράγοντα, αν μου επιτρέπετε, στην όλη διαδικασία αυτή. Αλλά το σημαντικό είναι ο άνθρωπος να έχει εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των αυτοκινούμενων οχημάτων. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε πολλά. Αυτά εισαγωγικά για την έκταση ίδιας πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βίμ Κύριε ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Η έκθεση αυτή δεν ασχολείται με το παρελθόν, αλλά θέλει να ανοίξει δρόμους για το μέλλον στην Ευρώπη. Όχι μόνο βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ως θεσμού, αλλά και για τους πολίτες και ο κύριος Φαντενκάμπ αναφέρθηκε στους πολίτες. Σε όσου ταξιδεύουν, για παράδειγμα με αεροπλάνα, με τρένα και οδικός. Προετοιμάζει την Ευρώπη για την εισαγωγή καινοτομιών. Καθήκον μας λοιπόν είναι να έχουμε πλήρη συνείδηση του ότι εκατοντάδες εκατομμύρια θα ταξιδέψουν ε, συνδρομικός, οδικός, αεροπορικός βεβαίως. Οπότε δουλειά μας είναι να δούμε πώς θα τους ε, παράσχουμε τις ε, βέλτιστες συνθήκες. Γι' αυτό καλωσορίζω την έκθεση αυτή του κυρίου ε, Φαντοκάμπ. Πολύ καλή έκθεση και από πλευράς της ομάδας μου. Έχουμε συνεργαστεί και διάφορα άλλα, διάφορες άλλες εκθέσεις και θα συνεργαστούμε στενά και για αυτή την έκθεση. Λοιπόν, το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και εξετάζει διάφορες μορφές μεταφορών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε εστιάσει κυρίως στα αυτόνομα οδικά οχήματα, αυτοκίνητα. Αλλά το θέμα ε, που τίθεται είναι ε, μήπως θα πρέπει να εξετάσουμε και την ε, αυτόνομη οδήγηση και οι άλλες μορφές μεταφορών. Για παράδειγμα, για τις, ε, την εσωτερική ναυσιπλοεία και την, ε, την πλοεία δηλαδή και ε, τις συνδρομικές μεταφορές. Βεβαίως αυτά τα θέματα θέτουν πολύ δυσχερείς προκλήσεις για όλους μας. Χρειαζόμαστε δηλαδή συστήματα που να είναι διασυνδεδεμένα, μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους ούτως ώστε να διασφαλίσουμε, μάλλον επιπλέον πρέπει να διασφαλίσουμε και την κυβερνοασφάλεια αυτών των συστημάτων και επίσης. Πρέπει και το να είναι προσαρμοσμένο ε, το κάθε σύστημα στις ανάγκες λειτουργίας του. Ως Ούγγρος μπορώ να σας ενημερώσω για τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε όταν χρειάστηκε να ε, περάσουμε από το πρώην Σοβιετικό σύστημα στο Ευρωπαϊκό σύστημα. Δεν είναι μόνο θέμα πλάτους για παράδειγμα των σεοδομικών γραμμών αλλά ε, για πολύ, πολύ ε, πιο προωθημένα αυτοματοποιημένα συστήματα που πρέπει οπωσδήποτε να είναι σωστά για να μην έχουμε τρομερά ατυχήματα. Είναι σωστή η προσέγγισή σας λέω καταλήγοντας κύριε Φαντεκάμπ. Αναφερθήκατε στην έρευνα και την ανάπτυξη που και αυτά είναι πολύ σημαντικά και ε, Συμφωνώ ότι πρέπει όλα αυτά να συμπεριληφθούν στον χρηματοδοτικό προγραμματισμό της περίοδου 21-27. Τώρα, πρέπει να υπάρξουν μεταβατικές περίοδοι για την εισαγωγή αυτών των νέων τεχνολογιών. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που ήδη ε, στις κάτω χώρες Έχετε ήδη κάνει τόσο πολλά για την οδική ασφάλεια και είστε στην πρωτοπορία. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε το αναγκαίο ε, δίκτυο ανεπτυγμένων τροπολογιών. Πέντε συνάδελφοι στείλαμε μία επιστολή στον ε, Επίτροπο που είναι αρμόδιος για τις μεταφορές στις αρχές του καλοκαιριού και ζητήσαμε να υπάρξουν νομοθετικές προτάσεις και οι επίτροποι μας απάντησαν αλλά δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα επίσης να τονιστεί η ανάγκη για περισσότερες νομοθετικές προτάσεις. Αλλά γενικά ευχαριστώ πολύ τον κύριο Φαντεκάμπ για τη συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Ιουλερή που αναφερθήκατε και, αυτήν, και σε αυτή την επιστολή την οποία και εγώ συνυπέγραψα γιατί θεωρώ ότι είναι ουσιώδη αυτά τα θέματα. Ο κύριος Λοτοσκι, Λοτόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον κύριο Φαντεκάμπ για αυτή την έκθεση. Η αυτοματοποιημένη κινητικότητα είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και ε, οι οδηγοί ε, το συζητούν πολύ γιατί θα σταματήσουν να οδηγούν. Συμφωνώ με την άποψη του συγητή από πολλές, για πολλά θέματα, αλλά θέλουμε να υπογραμμίσουμε τα θέματα. Πρώτα απ' όλα η ασφάλεια. Κατά τη γνώμη μου, η ασφάλεια πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα, οι ε, δοκιμές για τα ε, αυτόνομα οχήματα προχωρούν ε, πολύ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να μην υιοθετήσουμε τις σωστές διαδικασίες. Θυμάστε ότι έχουν υπάρξει ατυχήματα το θέμα δεν είναι ποιο θα ε, θέσει πρώτο στην αγορά ε, αυτόνομα οχήματα, αλλά ποιος ε, τελικά θα κερδίσει από αυτές τις νέες τεχνολογίες. Η ασφάλεια λοιπόν πρέπει να είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας και πρέπει να υπάρξει περισσότερη χρηματοδότηση των εργασιών προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, πρέπει να προειδοποιήσουμε όλους τους θεσμούς που εμπλέκονται για ορισμένους κινδύνους. Για παράδειγμα, να μην υπάρξει ενδεχόμενο τρομοκράτε να πάρουν τον έλεγχο οχημάτων. Επίση πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια για την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών. Να μην είναι αποκλειστικά θέμα των ε, μεγάλων επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να συνθλίψουν εντελώς τις μικρομεσαίες. Οι τεχνολογίες αυτές θα είναι φθηνέ, μόνο αν υπάρχει πλήρης πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα. Άρα η αγορά δεν θα πρέπει να κυριαρχείται από, τις, ε, από τους μεγάλους ομίλους επιχειρήσεων. Επίσης, ο ιδιοκτήτης ενός ε, οχήματος ε, αυτόνομης οδήγησης θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις διάφορες τεχνολογίες, στα ανταλλακτικά και όλα αυτά σε προσιτές τιμές. Και κάτι ακόμη. Πρέπει να ε, ασχοληθούμε και με τη μεταφορά εμπορευμάτων. Υπάρχουν ήδη αυτόματα μετρό, για παράδειγμα. Με βάση την πείρα από αυτές τις ε, πρόοδους, πρέπει να προωθήσουμε και την αυτόνομη μεταφορά εμπορευμάτων, λοιπόν. Και ε, την αυτόνομη οδήγηση σε άλλους τύπους μεταφορών. Επίσης, Πρέπει να ε, επενδύσουμε στις αναγκαίες υποδομές. Πρέπει να εξυγχρονιστούν οι υποδομές ε, στο δικό δίκτυο. Εάν δεν υπάρξει ε, η αναγκαία αυτή προσπάθεια εξυγχρονισμού, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά τα αυτόνομα οχήματα. Δεν πρέπει να υπάρξει τρομερή ανισότητα μεταξύ περιφερειών. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, σε μία περιφέρεια να μπορεί να υπάρξει πλήρης αυτόνομη οδήγηση και σε άλλη να είναι αδύνατο. Πρέπει λοιπόν να είναι και κερδοφόρος όλες αυτές οι τεχνολογίες. Ελπίζω να υπάρξει ε, θετική συνεργασία. Θέλω η έκθεση αυτή να είναι φιλόδοξη. Να λάβει υπόψη βέβαια ε, τα όρια, τα τεχνολογικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά να αξιοποιήσει όλε τι δυνατότητε που έχουμε ενώπιον μα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λοτόφσκι. Ο κύριο Φαν Μπίλτενμπεργκ από πλευρά τη Άλντε. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα συνεχίσω στα Ολλανδικά. Και... Νομίζω ότι είναι πραγματικά εξαιρετική αυτή η έκθεση πρωτοβουλία που κατέθεσε ο συνάδελφο. Όπω λέει και ο τίτλο, το θέμα είναι οι αυτοκινούμενε μεταφορέ, αλλά ο εισηγητή ε, ε, μου θυμίζει ε, ένα πρόγραμμα παλιό τηλεπτικό που είχαμε στην Ολλανδία για τις μεταφορές ε, στον αέρα και στους δρόμους και νομίζω ότι αυτό έκανε ο εισηγητής. Ε, το θέμα αυτό το επέκτηνε και όπως είπε είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα των αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων ε, το οποίο οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Μεγάλο λοιπόν ποσοστό και αυτό μπορούμε να το βελτιώσουμε στην Ευρώπη. Μπορούμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια μεταξύ άλλων αξιοποιώντας και τις τεχνολογικές εξελίξεις ε, των οχημάτων στο δρόμο. Πιο πολλέ λοιπόν αυτόνομε μετακινήσει, πιο πολλά αυτοκινούμενα οχήματα. Αυτό μπορεί να σημαίνει και πιο πολύ ασφάλεια, αλλά και πιο πολύ σωστή και ορθολογική χρήση και πιο λίγε εκπομπέ. Ε, όλα αυτά θα οδηγήσουν σε λιγότερε εκπομπέ διοξιδίου άνθρακα, γιατί πολύ απλά θα βελτιωθεί η κυκλοφορία θα υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό στόχος και επίσης θα ήθελα αυτό να τονιστεί πιο πολύ στην έκθεση γιατί υπάρχει μια παρανόηση κοιτώντα για παράδειγμα στην ε, παράγραφο 16 όπου μιλάμε για διάφορα προβλήματα στην κυκλοφορία τα οποία ενδεχομένω να προκληθούν από τα ξεκινούμενα οχήματα. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία αντίθετο. Τρία σημεία λοιπόν θα ήθελα να σημειώσω. Καταρχά, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια γενικότερα, είναι φατικό αυτό. Κατά δεύτερον, διαλειτουργικότητα, διαλειτουργικότητα τη τεχνολογία για να υπάρχει τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση και τρίτον προσέγγιση ενίσχυση της καινοτομία στην Ευρώπη και δύο μικρές παρατηρήσεις ε, στο τέλος καταρχάς για την ασφάλεια γενικότερα η γενικότερη ασφάλεια στην κυκλοφορία θα ήθελα να τονιστεί και η κυβερνοασφάλεια όμως είναι εντυπωσιακό το ότι το αναφέρει αυτό εισαγωγικά στα σχόλιά του Γιατί Δεν το βλέπω στην έκθεση όμως αυτό, γιατί είναι μπει κάπου στην έκθεση, γιατί βλέπουμε ότι και στην κινητικότητα υπάρχει κίνδυνος κυβερνοασφάλεια, χακαρίσματος. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρξει ασφάλεια για να υπάρξει και μεγαλύτερη αποδοχή των αυτοκινημένων οχημάτων στην Ευρώπη. Δεύτερο σημείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια εύρυθμα λειτουργούσα ευρωπαϊκή αγορά, οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται να είναι προσβάσιμες για όλα τα οχήματα, για όλους τους παραγωγούς. Και φυσικά ο καθένας έχει την ευθύνη του. Αλλά για μας ως νομοθέτες αυτό που είναι σημαντικό είναι να φροντίσουμε ότι θα υπάρχει διαλειτουργικότητα όλων των συστημάτων. Διαλειτουργικότητα λοιπόν. Αυτό θα ήθελα να τονιστεί πιο έντονα στην έκθεση. Όλα αυτά φυσικά χωρίς να διαταράξουμε και να στραβλώσουμε την ενιαία αγορά και την ελεύθερη αγορά. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα, αφορήσει, θα, θα μας, θα μας ε, επηρεάσει και την ε, νομοθεσία, το υποδομές. Τελευταίο θέμα. Καινοτομία. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και χαίρομαι που το αναφέρει ιδιαίτερα και ξεχωριστά ο εισηγητές και μιλάει και για ιδιαίτερους πόρους που θα αφιερωθούν στο θέμα αυτό από την Ευρώπη 2020 και πάρα πολύ σημαντικό είναι να προωθήσουμε την χαμηλότερη εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, γιατί αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να το τονίσουμε. Δύο μικρές παρατηρήσεις τώρα στο σημείο αυτό. Πρώτον, υπογραμμίζω και συμφωνώ απόλυτα αυτό που είπε ο εισηγητή για την κανόνα και τον κώδικα δεντολογία. Θα πρέπει να κάνουμε τέτοιε συζητήσεις δεντολογία για τέτοια σημαντικά θέματα που ανακύπτουν τα ζητήματα νέας τεχνολογίας, για παράδειγμα το data mining, τη τεχνολογία, πώς μπορούν να περιοριστούν από τον κώδικα δεντολογία. Χαίρομαι λοιπόν που κάνει αναφορά στην παράγραφο 15 στο θέμα αυτό, αλλά πιστεύω ότι οι παρατηρήσεις του για τα drones, για τα αυτοκίνημα αυτά οχήματα, ε, θα πρέπει να τονιστούν ιδιαιτέρους. Δεν μου φτάνουν αυτά που αναφέρει ο εισηγητής. Πώς λοιπόν θα ρυθμιστούν τα drones και στην έκθεση της πρωτοβουλίας της κυρίας Φώστερ σε μεγάλο βαθμό ε, επανέλθαμε στις βασικές αξιώσεις της ΕΑΣΑ ότι θα πρέπει να μην τεθούν μόνο απαιτήσει σε ό,τι αφορά το προϊόν αλλά και τη χρήση του προϊόντος των drones. Για παράδειγμα, ως επαγγελματίας, αν χρησιμοποιεί κανείς για παράδειγμα ένα drone ε, πάνω από ένα χωράφι, ε, θα πρέπει να ισχύουν διαφορετικές προδιαγραφέ. Αν για παράδειγμα, από το αν για παράδειγμα χρησιμοποιεί κανεί ένα ντρόουν με μια κάμερα για να βγάλει φωτογραφίε πάνω από ένα γήπεδο. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση η βασή αξιολόγηση κινδύνου θα επιτρέψει στην Ευρώπη να είναι καινοτομική σε ό,τι αφορά και θέματα ασφάλεια, χωρί όμω να κάνει υποχωρήσει σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλεια. Και ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση εδώ στο Κοινοβούλιο. Ακόμα και το κεφάλι του κυρίου Σιγητά, του κυρίου Μαρνέσκου, σε ό,τι αφορά τι προδιαγραφέ τη ΕΑΖΑ. Αλλά θα ήθελα να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε και τις ε, ε, πράξεις έτσι, κατανάθεση και θα πρέπει να αποφασίσουμε ποια είναι η ευρωπαϊκή αντίληψη και τι θέλουμε από ευρωπαϊκής άποψης να υποστηρίξουμε από πλευράς ασφάλειας, προκειμένου να τα αποδεχτούν όλοι τελικά αυτά. και σε οποιαδήποτε μόρφη μετακινήσεων και μεταφορών πάντα να επικρατεί ο παράγοντας της ασφάλειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαν Μίλτεμπεργκ για τα σχόλιά σας. Επόμενη ομιλήτρια θα είμαι εγώ γιατί είμαι συνεισηγήτρια. Κύριε Βιν Βαντεκάπ, ευχαριστούμε που μας αφυπνήσατε για αυτό το ζήτημα κέρια σημασίας με μεγάλες προσδοκίες ε, για την Ευρώπη. Το συζητά συνέχεια ο τύπος και δικαίως. Η αυτόνομη οδήγηση δεν συνιστάται σε μια απλή αλλαγή οχημάτων. Πρόκειται για μια βιομηχανική και πολιτιστική επανάσταση. Θα πάψουμε να είμαστε οδηγοί. Θα μετατραπούμε σε καταναλωτές, σε χρήστες ε, οχημάτων στο μέλλον. Αυτό θα αλλάξει και τις συμπεριφορές μας. Και θα γεννήσει και νέες. Γι' αυτό κύριε Βιμ Βαντεκάμπ, ε, εδώ καθώς τελειώνει η θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε την ευκαιρία να ε, ορίσουμε έναν ορίζοντα και ένα πλαίσιο. Αυτό είναι στόχος της Επιτροπής μας πριν από το τέλος της θητείας μας. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι τα οχήματα αυτά και ξεκινάω από το αυτόνομο αυτοκίνητο για το οποίο συζητούν απαντές ε, θα πρέπει να βασιστούν ε, στους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις επενδύσεις, στην έρευνα, στην καινοτομία, στην γενετικότητα των μεταφορών, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε ότι αυτό που θα πρέπει να μας ανησυχεί πρωτίστως είναι ο περιβαλλοντικός στόχος. Σε περιβαλλοντικά θέματα, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, σήμερα γνωρίζουμε ότι κάθε αυτοκίνητο χρησιμοποιείται 5% ε, του χρόνου της. Δηλαδή το 95% του χρόνου του τι κάνει το αυτοκίνητο. Κοιμάται σε ένα πάρκινγκ μπροστά μας. Μένει ακίνητο. Αχρησιμοποιητό. Αλλά σε αυτό το χρόνο που παραμένει χρησιμοποιητό μας κοστίζει χρήματα διότι κάθε Ευρωπαίος πολίτης δαπανά μεταξύ 5 και 6.000 ευρώ μόνο για τη συντήρηση ενός αυτοκινήτου το οποίο τον περισσότερο χρόνο κοιμάται. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια ευρώ που σπαταλώνται άσκοπα. Τα αυτοκίνητα αυτά καταλαμβάνουν και χώρο και μας κοστίζουν χρήματα. Αλλά προσοχή. Το θέμα που ανακύπτει από όλα αυτά είναι ότι θα πρέπει να έχουμε σωστά ε, αντίδραση ως άνθρωποι που ζούμε στον 21ο αιώνα. Μιλάμε για μείωση του στόλου των αυτοκινήτων και της κατανάλωσης ενέργειας. Όχι το αντίθετο. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Μας λένε ότι το 90% των ατυχημάτων οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα και ότι η αυτόνομη οδήγηση θα βοηθήσει στη μείωση της νησιμότητας και του αριθμού των ατυχημάτων. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο διακύβευμα. Κύριε Βαν Μίτελμπεργκ, ε, αναφερθήκατε και στο συγκεκριμένο ζήτημα της ασφάλειας των drones. Κάτι πολύ δύσκολο. Ανεξάρτητα από τους εμπορικούς στόλους, ε, σήμερα ήδη έχουμε τέτοια πειράματα. Μιλάμε για drone ψυχαγωγικά που ε, όλο και περισσότερο συναντάμε. Τίθενται ζητήματα και επιδόσεων αλλά και ασφάλειας. Και εκεί λοιπόν προκύπτουν ε, προκύπτει ότι η κατεξοδότηση πράξης για τα θέματα αυτά δεν, αφορούν, δεν εξετάζουν όλα τα ζητήματα τη τεχνητή νοημοσύνη και τη συμπεριφορά των drones. Χρειαζόμαστε λοιπόν συγκεκριμένε συστάσει επί του ζητήματο στην έκθεση αυτή. Κύριε Βίμ Βαντεκάμπ, ε, αναφερθήκατε στην αναγκαιότητα για μια νομοθεσία και ειδικότερα για τα δεδομένα. Αλλά κυρίω στην παράγραφο 8 λέτε ότι πρέπει να έρθουν όλα τα εμπόδια χρήση δεδομένων. Πρέπει να διευκρινίσουμε ποια είναι τα εμπόδια αυτά και ποιο θα πρέπει να μπορεί να τα χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα. Οι κατασκευαστές, οι καταναλωτές, όλα αυτά τα ερωτήματα πρέπει να τεθούν αυτή τη στιγμή. Σήμερα πάρα πολλοί οργανισμοί διεξάγουν διάφορες εκστρατείες. Ε, ε, είδα έγινε μια εκστρατεία για τη ε, δημοσιοποίηση των δεδομένων που υπάρχουν στα αυτοκίνητα ώστε να έχουν πλήρη έλεγχο οι χρήστες Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω ότι εδώ ήταν πολύ άριθμοι ε, οι βουλευτές από πολλές ε, πολιτικές ομάδες που έγραψαν στην Κομισιόν και απέτησαν νομοθεσία ευνοϊκή για τους καταναλωτές ε, περισσότερο από ότι για τους κατασκευαστές. Και ελπίζω να εγκριθούν και οι τροπολογίες που θα προτείνω εγώ για αυτή την έκθεση προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι δεν αναφέρεστε επαρκώ στην τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Βαντεκάμπ, στην εκθεσή σα. Οι αλγόριθμοι που θα επεξεργάζονται και θα βελτιστοποιούν τα δεδομένα θα πρέπει να υποβάλλονται σε έναν ε, κώδικα διοντολογία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, ώστε να επιτηρείται η, η καλή χρήση των δεδομένων αυτών. Εκεί θα πρέπει να παίξει το ρόλο το διαιτητικό που έχει η Ευρώπη η οποία δεν έχει δράσει επαρκώς προληπτικά όσον αφορά τα δεδομένα που αφορούν τους ρήπους. Ξέρουμε με τι θα κυκλοφορούν αυτά τα μελλοντικά οχήματα μέσα μεταφοράς. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Εκεί τίθε το ενεργειακό ζήτημα, κύριε Βαντεκάμπ, και το ζήτημα των υποδομών. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Βαντεκάμπ. Ένα αυτονόμο αυτοκίνητο Ξέρετε, για να ανοιχνεύσει ε, μια λιμνούλα από νερό, ένα λάκκο από νερό, μικρό, χρειάζεται πάνω από 18 δισεκατομμύρια ε, στοιχεία δεδομένα το δευτερόλεπτο για να ανοιχνεύσει μια, μια μικρή λακκούβα με νερό. Αντιλαμβάνεστε τι θα καταναλώνει ενεργειακά για να μπορέσει να σκεφτεί έτσι ως αυτόνομο όχημα ότι πρόκειται για μια λακκούβα. Μιλάμε για τεράστιες υποδομές ε, και για ε, το ζήτημα των data center. Τα data center αυτά πού θα βρίσκονται για να ε, λειτουργεί αυτό το αυτόνομο όχημα, πού θα τα βάλουμε, ποιος θα τα χρηματοδοτήσει, πώς θα κοστίσουν αυτά τα data center, θα λειτουργούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό ελπίζω και εγώ. Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τεθούν τώρα ως ερωτήματα. Ε, όλα τα θέματα αυτά των υποδομών, διότι εάν φυσικά δεν δημιουργήσουμε τις απαραίτητες υποδομές, ε, δεν θα λειτουργήσει το όλο εγχείρημα. Επίσης, κύριε Βιμβαντεκάμπ, θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπενθυμίσουμε ένα πράγμα. Τα όσα θα δούμε μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια και εμείς και η αυτοκινητοβιομηχανία δεν έχουν να κάνουν καθόλου με όσα είδαμε τα τελευταία 50 χρόνια. Μιλάμε για μια επανάσταση στην απασχόληση. Μιλάμε για μια βιομηχανία που απαριθμεί 12 εκατομμύρια θέσεις εργασία. Χωρίς να μιλώ για τους παρατραχάμενους, τι θα γίνει με αυτές τις θέσει εργασία, με αυτούς τους μισθωτού οι οποίοι σήμερα βλέπουν τα κράτη να λένε θα εγκαταλείψουμε τις ορεικτές πηγές ενέργειας, θα επενδύσουμε στις νέες πηγές ενέργειας. Χρειάζεται και ένα σχέδιο ε, ε, επανεκπαίδευσης αυτών των ανθρώπων. Εκεί θα πρέπει να γίνουν κάποιες επενδύσεις. Ε, να σας υπενθυμίσω ότι αύριο το αυτοκίνητο δεν θα είναι πια ατομική περιουσία, θα είναι κοινή περιουσία. Πώ θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτή την κινητικότητα που θα είναι επιμερισμένη, που θα είναι κοινή κινητικότητα, γιατί έχετε δίκαιο, κύριε Βαντεκάμπ, όταν αναφέρεστε στην ατμοσφαιρική ρήπανση και λέτε τι θα κάνουμε με όλη αυτή τη συμφόρηση. Θα πρέπει λοιπόν να περάσουμε από την ατομική στην κοινή κινητικότητα μέσα στον 21ο αιώνα. Και το στίχημα είναι τι θα γίνει με τις επενδύσεις, πώς εμείς η Ευρώπη μέσω των επενδύσεων θα καταφέρουμε να ξεκινήσουμε νέες αλυσίδες παραγωγής και να υλοποιήσουμε τις μεταφορές του αύριο. Και εκεί έχουμε ένα πρόβλημα βασικό. Διότι δεν έχουμε κάνει τίποτα σχεδόν. Έχουμε καθυστερήσει ως Ευρώπη. Δεν λέω ότι έχουμε καθυστερήσει υπερβολικά, αλλά έχουμε καθυστερήσει. Τώρα θα πρέπει να κινηθούμε με τους νέους παραγόντες της startup, ε, τις οποίες υποστηρίζουμε και εμείς στην Επιτροπή μας, αλλά θα πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να ξαναβρούμε την ηγετική μας θέση ως Ευρωπαίοι. Εκεί είναι η δυσκολία, διότι η Κίνα δεν μας περιμένει, ούτε οι Πολιτείες μας περιμένουν. Αλλά και οι τρόποι κινητικότητας που θα επέλθουν δεν θα μας περιμένουν. Αυτά ήθελα να πω για να συμβάλλω στην εκθέση σας κύριε Βιμβαντεκάμπ. Κύριε Κορ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δήμ, σε ευχαριστώ. Πολύ καλή έκθεση πρωτοβουλία. Ένα σημείο θα αναφέρω. Η προετοιμασία των ανθρώπων για να μπορέσουν να αποφελθούν ε, από αυτές τις νέες τεχνολογίες. Ε, η τεχνολογία προχωρεί και πολλά δεν τα θέλουν οι άνθρωποι και δεν τα αποδέχονται. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να αναφέρουμε στην έκθεση ότι πρέπει τα συστήματα Βοήθηση προ την οδήγηση θα πρέπει να βοηθήσουν για την αποδοχή αυτή τη τεχνολογία. Είναι προϋπόθεση για να καταλήξουμε στα αυτόνομα οχήματα. Να είναι ε, λοιπόν ένα βήμα η ε, εισαγωγή συστημάτων βοήθεια στην οδήγηση. Δεν μπορούμε να, το, ε, να μην περάσουμε μέσα από αυτήν την ενδιάμεση κατάσταση. Η κυρία Ντεμόντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους άλλους ε, σκιώδεις για την ε, συμβολή τους. Όπως υπόθηκε, το μέλλον ανήκει στα αυτόνομα οχήματα. Θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο όχι βέβαια μόνο τα ε, αλλά και πολλά άλλα οχήματα. Και επίσης ε, τα επιβοηθητικά συστήματα για την οδήγηση των φορτηγών μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Στην Ιταλία είχαμε σοβαρά οδικά ατυχήματα, για παράδειγμα κάποια φορτηγά που μετέφεραν ε, έφλεκτα υλικά. Και αυτό πρέπει λοιπόν να το κοιτάξουμε. Δεν είναι μόνο θέμα λοιπόν ε, αντιμετώπισης αλλά και αποφυγή αυτών των ε, δυστυχημάτων. Και φυσικά πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα των ε, άλλων μορφών μεταφορών. Και θα έχει φυσικά επιπτώσει και στην απασχόληση το θέμα αυτό. Πολλέ ε, θέσει εργασία θα χαθούν. Γιατί ξέρετε ότι το μέσο των μεταφορών απασχολεί πολλού εργαζόμενου και από περιβαλλοντική άποψη. Βεβαίω, όπω είπατε και εσείς, κυρία Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν τα οχήματα να χρησιμοποιούνται τόσο μικρό ποσοστό του χρόνου. Ενώ παράλληλα έχουμε προβλήματα κυκλοφοριακής συγχώρησης. Συμφόρησης. Γιατί ένα μεγάλο τμήμα της επιφάνειας των πόλεων μας και των οικοδομών μας χρησιμοποιούνται για να παρκάρουν και να κυκλοφορούν τα οχήματα. Και επίσης αυτό δημιουργεί και η κυκλοφορία δηλαδή, των οχημάτων δημιουργεί πολλά προβλήματα στους πεζούς για να μπορούν να κυκλοφορούν άντα στις πόλεις. Τα έχουμε αναφέρει αυτά επανειλημμένα. Καθίσταται λοιπόν δυνατόν να δημιουργήσουμε τις ε, σωστά αποδοτικές υποδομές στον τομέα αυτό. Αλλά αυτό θα έχει φυσικά το κόστος του. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε υπόψη μας και να καθορίσουμε ποιος θα πληρώσει για τις υποδομές. Ποιος θα πληρώσει για την εισαγωγή αυτών των αυτονόμων οχημάτων. Επίσης ε, πρέπει να έχουμε υπόψη και την ε, αλυσίδα υπετιότητας και ευθύνης. Δεν είναι μόνο θέμα ε, παραβίασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχει θέμα ποινική ευθύνης, υπάρχει θέμα αστικής ευθύνης αν θέλουμε λοιπόν να τα καλύψουμε όλα αυτά από την αρχή μέχρι το τέλος, τότε πρέπει να εμπλέξουμε και όλες ε, τις ε, επιχειρήσεις που εμπλέκονται, όχι μόνο τα άτομα. Και τέλος, ε, η προστασία του ιδιωτικού βίου θα παίξει ρόλο κλειδί. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Όταν συζητήσαμε τα θέματα ασφαλούς πρόσβαση στα δεδομένα. Είναι λοιπόν γενικά περίπλοκο το θέμα αυτό. Γι' αυτό πρέπει να καθορίσουμε σωστά τις λεπτομέρειες, αλλά να καλύψουμε και γενικότερα το ευρύ φάσμα. Ο κύριος Έρτουγκ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα και σε εσά. Να ευχαριστήσω και εγώ τον συνάδελφο τον κύριο Φοντενκάμ για την έκθεση του. η επικοινωνία στο βαθμό που το κρίνω εγώ, θεωρώ ότι περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία αφορούν τους ε, αυτοκινητοβιομηχανούς και το θέμα λοιπόν της ασφάλειας, το θέμα της αστικής ευθύνης, το θέμα της προστασίας των δεδομένων και της πρόσβασης των δεδομένων κυβερνού ασφάλεια, ε, συνδεσιμότητα και ε, αποδοχή από πλευρά τη κοινωνία τη τεχνολογία και φυσικά οι επιπτώσει στην αγορά εργασία. Να αναφέρω ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία είτε πρόκειται για τους βιομηχάνες, είτε πρόκειται για τους ε, προμηθευτές, θα πρέπει να κάτσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και αυτό θέλω να μεταφέρω και στους συναδέλφους, ότι θα πρέπει να, να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους ε, προμηθευτές. Εδώ λοιπόν ε, πραγματικά έχουμε να επενέσουμε αυτά που έχουν γίνει. Εγώ δεν τα παρουσιάζω όλα Ρόδινα, αλλά στην ε, περίπτωση αυτή θεωρώ ότι η βιομηχανία έχει διακρίνει τα σημεία της ε, εποχής μας αυτής και έχει προετοιμαστεί. Τώρα, να αναφέρω το σημείο 1, το οποίο ε, ανέφερα και προηγουμένω. Το θέμα λοιπόν της συνέπειας. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένα μέτρα. Αυτό ακούμε και από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, ότι μπορούν να αξιοποιήσουν ήδη τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά λείπει το νομοθετικό πλαίσιο. Αυτή η ρύθμιση η οποία πρέπει να υπάρχει. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτήν. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη. Αυτή πρέπει να κάνει την πρώτη, το πρώτο βήμα. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την έγκριση τέτοιων ε, οχημάτων, θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς ε, προδιαγραφές και για τα θέματα ασφάλειας προφανώς, αλλά και για άλλα ζητήματα όπως για παράδειγμα οι Αυτόνομη και μη διαδικτυωμένη ε, οδήγηση ονομάζεται. Όταν μιλάμε για δικτύωση, ξέρουμε ότι υπάρχει δικτύωση μεταξύ των οχημάτων και του περίγυρου. υποτομές και ούτω καθεξής. Αυτό είναι απόλυτο ως απέτηση προκειμένου να υπάρχει αυτονομία οδόγηση και προκειμένου να κινηθούμε και να εξελιχθούμε μέχρι την πλήρη αυτοματοποίηση σε ό,τι αφορά την προστασία δεδομένων τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι προφανώ πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό και πάρα πολύ ευαίσθητο, ακαθόδε. Θα πρέπει λοιπόν να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα. Ποιο θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα επί τη αρχή, σε πού θα αποθηκεύονται τα δεδομένα, ποιο θα τα αποθηκεύει, και ποιος ε, έχει δικαίωμα να τα διαχειρίζεται στη συνέχεια αυτά τα δεδομένα, να τα χορηγεί σε τρίτους και το καθεξής. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν ε, θέλουν απαραίτητα να δώσουν ε, τα δικαιώματα αυτά. Ενδεχομένως όμως και άλλες τεχνολογική άλλα άλλε βιομηχανίε να έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και να μην χρειάζεται να τα πληρώνουν. Αυτό θεωρώ ότι είναι λογικό και εύλογο. Και επίση αυτό δεν μπορεί να είναι σε αποκλειστικά εθνική αρμοδιότητα ως θέμα, πιστεύω. Θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα γιατί οι τεχνολογίες αυτές, αυτή η αλλαγή νοτροπία αν θέλεις, Καρίμα, όπως την ανέφερα, δεν μπορεί να γίνει σε εθνικό μόνο επίπεδο. Θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό, μη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα αυτό και να το βάλουμε τι προδιαγραφέ. Επίση, αύξηση τη αποτελεσματικότητα, τη αποδοτικότητα. Πολύ καλό ο στόχο σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία, αλλά παράλληλα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι με τις τεχνολογίες αυτές ενδεχομένως να καταλήξουμε να έχουμε πιο πολλή κυκλοφορία τελικά. Και άρα ό,τι κερδίσουμε από την αύξηση της αποτελεσματικότητας να το χάσουμε γιατί θα υπάρχει μεγαλύτερη κυκλοφορία και άρα μεγαλύτερα αποτελιαρίσματα και μεγαλύτερη συμφόρηση γενικότερα. Να το σκεφτούμε λοιπόν αυτό. Και τέλος, πιστεύω ότι η, έκθεση ε, καλά κάνει και δεν επικεντρώνεται μόνο στις οδικές μεταφορές και την αυτόνομη οδήγηση στις ε, οδικές μεταφορές. Ε, περιλαμβάνονται και οι άλλοι τομείς όπως για παράδειγμα η αεροπορία και η ναυσιπλοεία και αυτό είναι απαραίτητο αν θέλουμε πραγματικά να υπάρχει σωστή ε, κυκλοφορία ε, με ροή. Και η συνδραδρομή λοιπόν είναι πολύ απαραίτητη και εγώ δεν θέλω να κάνω ε, διαφήμιση για την ε, πατρίδα μου, την προσωπική μου πατρίδα, αλλά στο 2007-2008 ήδη είχαμε στην Ευέργη μια πλήρως αυτοματοποιημένη ε, ένα σύστημα σιδηροδρόμων και τρένων μέσα στην πόλη. Και αυτό νομίζω ότι αύξησε την αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ. Και τώρα να ακούσουμε τον επόμενο μιλητή. Ο κύριος Λούντγκριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μόνο που τα ακούω αυτά, μου σηκώνονται η τρίχα ορθιά. Για μένα τα αυτοκίνητα είναι έργα τέχνης. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αγοράσω ένα αυτοκίνητο το οποίο θα οδηγεί στη θέση μου. Κάνω και ράλι, κάνω και, και τέτοια ράλι. Είμαι λάτρης της ταχύτητας, 200 χιλιόμετρα στα βάση μας. Και θεωρώ λοιπόν ότι και η αυτοκινητοβιομηχανία ε, έχει βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν πρόκειται λοιπόν να δεχτώ ποτέ ένα αυτοκινούμενο όχημα να αποφασίζει το όχημα για μένα. Εντάξει, ενδεχομένω ε, ένα ταξί μέσα στην πόλη είναι άλλο θέμα. Αλλά τώρα να είμαι στο δάσο και να χιονίζει και να μην έχω τον έλεγχο του οχήματο, για παράδειγμα, ένα φορτηγό να μην έχει οδηγό άνθρωπο, πώ θα να εξελιχθούν όλα αυτά. Στις πόλεις ενδεχομένω να λειτουργήσει ο σύστημα αυτό, αλλά στην Ήπεθρο αυτό δεν πρόκειται ποτέ να περάσει ως ε, σύστημα και εγώ ποτέ δεν ε, πρόκειται να δεχτώ ένα τέτοιο σύστημα, γιατί εγώ θέλω να οδηγώ το αυτοκίνητο και όχι αυτό το αυτοκίνητο να με πηγαίνει εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ρενγκρένα. Ε, ακούσαμε καθαρά το μήνυμά σα. Αλλά αποφύγετε τα 200 χιλιόμετρα την ώρα με στο δάσο. Είναι θέμα ασφάλεια. Κυρία Γιάλα Σέντερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Φαντεκάμπ για τα συμπαθητικά του λόγια. Νομίζω ότι το θέμα αυτό μας θέτει ενώπιον των ε, αμέσων ευθυνών μας γιατί ήδη εταιρείε ε, όπως η Tesla και άλλες στη Silicon Valley, αλλά ακόμη και στην Ευρώπη κάποιες εταιρείε προωθούν ε, αυτή την αυτόνομη οδήγηση και στην Ανατολική Ασία. Να θυμίσω ότι το πρώτο μετρό χωρίς οδηγό ήταν στον Detroit στις αρχές δεκαετίας του 1990. Ήταν ε, ένα αέριο. Αλλά το Detroit ήταν ήδη σε κατάσταση κατάρρευσης, είχαν κλείσει αυτοκινοβιομηχανίες, ε, οι υποδομές ήταν άθλιες, υπήρχε τεράστια ανεργία και ανασφάλεια. Και ήταν ένα, ε, υπήρχε ένα πρόγραμμα για να βγει από αυτή την κατάσταση, αλλά το μετρό ήταν καταπληκτικό και θαυμάσιο. Οπότε ρωτώ κύριε Φαντεκάμπ, θαυμάσιο το κείμενό σας που αναφέρεται στη σχέση μεταξύ της αυτόνομης οδήγησης και του ατόμου, είτε είναι αεροπλάνο ή καράβι, αλλά δεν αναφέρεται επαρκώς στην, ε, στις υποδομές. Και το είδαμε και στην Silicon Valley για την περίπτωση της Tesla, ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Γιατί ε, βεβαίως η αυτόνομη οδήγηση δεν γίνεται στο διάστημα. Ακόμη και εκεί υπάρχουν βέβαια τα διαστημικά απορρίμματα. Αλλά ε, στη γη υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχει η, η σήμανση. Ε, το θέμα είναι τι θα γίνει, ποια είναι η άσφαλτος ε, επί των οποίων θα κινείται, ποιε είναι οι είσοδοι και οι έξοδοι από τις πόλεις. Και επειδή το κείμενό σας ε, αναφέρεται για την ασφάλεια και για τις υποδομές, όπου το θέμα είναι να υπάρξει σωστά νομοθετική ρύθμιση όλων αυτών, αυτό που πρέπει λοιπόν να δούμε είναι πώς θα αναφερθούμε σωστά στις προϋποθέσεις για την αυτόνομη οδήγηση. Πώς θα βελτιώσουμε την ασφάλεια, πώς θα υπάρξουν οι αναγκαίοι κανόνες για τις υποδομές και την ασφάλεια και για τις επενδύσεις. Μπορεί να φτιάξουμε τα καλύτερα αυτόνομα ε, οχήματα στην Ευρώπη, αλλά μπορεί να καταρρεύσει η γέφυρα Μοράντι όταν θα περνάνε. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές. Πριν επενδύσουμε σε αυτά τα θαυμάσια συστήματα, με τα οποία συμφωνώ απόλυτα, και είναι πολύ καλό, για παράδειγμα, οι ηλικιωμένοι να μην χρειάζεται να οδηγούν, να μπαίνουν σε αυτόνομα οχήματα και έτσι να έχουμε περισσότερη ασφάλεια. Πρέπει να γίνουν αναγκαίε επενδύσει. Και για τα δεδομένα, βεβαίω συμφωνώ, κυρία Πρόεδρε, με αυτά που είπατε, είναι θεμελιώδε. Είδαμε ότι η Τέσλα υπογράφει ε, συμβάσεις με τους ε, αγοραστές των οχημάτων της. Αλλά πρέπει να υπάρξει δημόσια ρύθμιση, να μπορεί να γίνεται η αναγκαία έρευνα, γιατί αυτά, αυτά τα αυτόνομα συστήματα θα είναι το πετρέλαιο του 21ου αιώνα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει δημόσιος έλεγχος. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε στρέφουμε και πάλι, όχι μάλλον στρέφουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Κλέρ Ντουπρέ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Α, όχι, δεν είστε εσεί. Κλέρ Ντουπρέ. Ωραία, και για τι δύο σα παρακαλώ το πολύ τέσσερα λεπτά. Ο χρόνο μετράει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την έκθεση και για τη συζήτηση που προσθέτει ε, πολλά στη συζήτησή μας. Λοιπόν, έχω μόνο τέσσερα λεπτά. Δεν ξέρω αν θα με φτάσουν. Θα ασχοληθώ με τα πιο σημαντικά. Πρώτον, ευχαριστούμε την Επιτροπή σα που θέτει το θέμα τη αυτόνομη οδήγηση. Και ελπίζω ότι θα είναι απλώ η αρχή του διαλόγου και για θέματα ουσία, που είναι διάφορα και δυσχερή, αλλά και για τα συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα. Όλοι καλέσατε να υπάρξει νομοθεσία. Και βεβαίω θα υποβάλουμε νομοθετικέ προτάσει. Οπότε θα ασχοληθείτε και με συγκεκριμένα νομοθετήματα με συγκεκριμένου κανόνε. άρα είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η συζήτηση. Η έκθεσή σα ασχολείται με πάρα πολλά θέματα. Πολλά που έχουν να κάνουν με την αυτόνομη οδήγηση, ασφάλεια, ψηφιοποίηση, θέματα διοντολογία, κοινωνικά θέματα, θέσεις εργασία και την υποδομή που αναφέρθηκε. Αλλά θέτει επίση. και θέματα διαφόρων ε, μοδο, ε, ειδών μεταφορών. Για παράδειγμα, ε, ποταμοπλοεία, αεροπορία. Βεβαίω εστιάζεται στι οδικέ μεταφορέ, αλλά υπάρχουν προκλήσει και για άλλα είδη μεταφορών. Λοιπόν, να ασχοληθώ με ορισμένα από τα θέματα που και εμεί θεωρούμε πολύ σημαντικά για τι οδικέ μεταφορέ. Θέματα που αναφέρατε. Νομίζω ότι συμφωνείτε ότι η ανακοίνωση του Μαΐου είναι πολύ ευρεία. Εστιάζει στα οχήματα και το οδικό δίκτυο, αλλά αντιμετωπίζει, μάλλον αναφέρει, πολύ ευρύτερα προβλήματα. Γιατί εστιάσαμε στις οδικές μεταφορές. Γιατί ε, πήγει το θέμα αυτό. Πρέπει να δείξουμε στον έξω κόσμο ότι η Ένωση έχει το δικό της πρόγραμμα αυτόνομης οδήγησης, ότι δεν έχει απλώς ε, ε, την πρόθεση να κάνει πολιτικές διακηρύξεις, αλλά ότι θέλει να θέσει πρωτοβουλίες, για, ε, πρωτο, συγγνώμη, προτεραιότητες για την έρευνα, τις υποδομές κτλ. Είμαστε το πρώτο μπλοκ παγκοσμίω που έχει θέσει το θέμα γενικά της αυτόνομης οδήγησης, τώρα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την ασφάλεια. Αναφερθήκατε στην κυβέρνηση ασφάλεια και την πρόληψη των ατυχημάτων. Τονίζω ότι στα πλαίσια του UNICE, όπως λέει και η έκθεση, αλλά και στην Ένωση, εδώ και πολύ καιρό έχουμε αρχίσει να εκπονούμε διάφορους κανονισμούς για την κυβερνοασφάλεια των οχημάτων και θα καταλήξουμε σε κάποια πρώτα βήματα τέλος του χρόνου και κατόπιν θα προτείνουμε νομοθετήματα. Γίνεται λοιπόν παγκοσμίω. Γιατί λέω παγκοσμίω, Γιατί η αυτόνομη οδήγηση είναι παγκόσμιο θέμα. Αλλά άρα είναι προ το συμφέρον όλων μα να υπάρξουν παγκόσμιες προδιαγραφές. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι χάρη στην πίεση της Κομισιόν το UNICE έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας για την αυτόνομη οδήγηση. Λοιπόν, ε, προπαρευόμεθα για το θέμα αυτό. Για την ασφάλεια. Η Επιτροπή σας θα εξετάσει τον κανονισμό γενικής ασφάλειας που εγκρίθηκε τον περασμένο Μάιο που δεν ασχολείται, δεν μόνο με συμβατικά θέματα ασφάλεια αλλά ανοίγει το δρόμο και για την αυτόνομη οδήγηση. Συγκεκριμένα μέτρα προβλέπονται για την αυτόνομη οδήγηση. Γι' αυτό σας ε, ενθαρρύνουμε να ασχοληθείτε ταχαίως με αυτόν τον κανονισμό. Αναφερθήκατε με την ε, καταγραφή των ε, δεδομένων των οχημάτων. Βεβαίως ο κανονισμός το αναφέρει για να καθοριστούν τα θέματα υπετιότητας μεταξύ της μηχανής και ε, του οδηγού. Για τα θέματα διοντολογίας και κοινωνικής αποδοχής. Προτιθέμεθα να δημιουργήσουμε ένα φόρουμ που θα ασχοληθεί με τα θέματα διοντολογίας της αυτόνομης οδήγηση. Ελπίζουμε να αρχίσει να λειτουργεί πριν από το τέλος του χρόνου. Και σταματάω λοιπόν εδώ. Θα δώσω το λόγο στην Κλέα. Έχετε ένα λεπτό κυρία Ντεπρέ. Πολύ σύντομα. Η έκθεσή σας ασχολείται με πολλά θέματα. Καλύπτει όλες τις μορφές μεταφορών. Όλους τους τρόπους μεταφορών. Δεν ασχολούμεθα μόνο με τις οδικές μεταφορές. Ασχολούμεθα με όλους. Βεβαίως ε, για κάθε μορφή μεταφορών ασχολούμεθα διαφορετικά και είμαστε σε άλλο επίπεδο. Για παράδειγμα για την ε, ποταμοπλοεία ασχολούμεθα διεθνώ και στον αεροπορικό τομέα επίσης υπάρχει πρόοδος επί συγκεκριμένων κανόνων Ορισμένοι ανεφερθήκατε στη σύνδεση με την τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαίως είμαστε σε αρχικό στάδιο ακόμη πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα τι επιπτώσεις θα έχει η εισαγωγή ε, αυτού του τρόπου μεταφορών. Αυτό ισχύει για ε, όλες τις μορφές μεταφορών. Θέλουμε να μας βοηθήσετε λοιπόν για να συνδεθεί στενότερα η έρευνα και η καινοτομία με την ε, νομοθεσία. Και ελπίζω να μπορέσετε να βοηθήσετε την Κομισιόν σε αυτό. Εξετάζουμε την κινητικότητα, την επίπτωσή της ε, στην κατάσταση της πόλης. Θέλουμε να υπάρξουν ε, προγράμματα βιώσιμης κινητικότητας για να λάβουν και οι πόλεις ε, τις ευθύνες τους. Να εμπλακούν σε αυτή την προσπάθεια και να την λάβουν υπόψη τις απαιτήσεις του τομέα αυτού στην πολεοδομία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντουπρέ. Να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για την έκθεση αυτή είναι η 12η Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Αλλά φυσικά δεν μπορούμε να κλείσουμε χωρίς τον εισηγητή, οπότε δίνω το λόγο στον κύριο Βιν Βαντεκάμπ. Φοβηθήκατε ε, για λίγο. Ε, Πρόεδρε, εγώ δεν φοβάμαι ποτέ. Και για να είμαι ξεκάθαρος. Είπατε οι τροπολογίες ε, θα πρέπει να κατατεθούν 2 Σεπτεμβρίου. 12 Σεπτεμβρίου. 12 Σεπτεμβρίου βλέπω όμως όχι. Δεν ξέρω. Αν θέλετε να μου το επιβεβαιώσετε παρακαλώ. 12, 12 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Καταρχάς, Πρόεδρε, λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η DG Growth και η DG Move μα απέφτυναν το λόγο. Πολύ καλό συνδυασμό. πάντα. Δύο γενικοί διευθυντέ. Γενικέ γενικές διευθυντρίες. Όχι μόνο καλό συνδυασμό, αλλά και μεγάλη πρόκληση πάντα. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για όλες τις παρατηρήσεις. Ε, ο Μάρτιν Φούξ σημειώνει από την Επιτροπή, από την Γραμματεία της ε, Επιτροπή και τις ε, ασχόλια του Τόμας, του κυρίου Φαν Μίλτερ που έχει, του κυρίου Ερτούκ. Θεωρώ ότι περιλαμβάνουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα κληθούμε να τα συζητήσουμε τις επόμενες εβδομάδες και τις παρατηρήσεις του κυρίου Κόχ για την επόμενη την ε, μεταβατική φάση, την ενδιάμεση φάση των συστημάτων ε, μεταφορών θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ εύστοχε και πραγματικά επεσήμεναν πάρα πολύ ε, σωστά στοιχεία. Και η κυρία Φαμίλτεμπεργκ, όντω ε, μίλησα κι εγώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις πράξεις κατεξουσιοδότηση και την άθεση για τα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη για τα drones. Περίμενα λοιπόν τις τροπολογίε σα με ανυπομονησία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξέρει ότι οποιαδήποτε στιγμή θέλει να έρθει να πιούμε ένα καφέ για να συζητήσουμε πιο πολλές λεπτομέρειες είναι ευπρόσδεκτη. Αυτό που συγκρατώ είναι η παρατήρηση του κυρίου Ερτούγκ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συνοδεύσει όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίε από νομοθετική άποψη προκειμένου να δημιουργηθεί το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο που χρειάζεται. Αυτό να το σκεφτούμε, γιατί δεν μπορούμε φυσικά να υποχρεώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση νομοθεσία για τεχνολογία η οποία ακόμα δεν υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε να εμποδίσουμε και την ευρωπαϊκή βιομηχανία από το να αναπτυχθεί με ευρωπαϊκή προσέγγιση. Αυτό ε, νομοθέτη ενδιαφέρει ιδιαίτερα και σίγουρα θα το σκεφτούμε τις επόμενες εβδομάδες. Χαίρομαι, κυρία Πρόεδρε, που προασπίζετε τα δικαιώματα των εργοδοτών στην αυτοκινητοβιομηχανία. Πρώτη φορά. Δεν το έχουμε ακούσει αυτό πολλές φορές από πράσινο. Πολιτικό. Να προασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία. Μεγάλη πρόοδος λοιπόν αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και παρακαλώ να συνεχίσετε και εσείς να σκέφτεστε μαζί μου προκειμένου να εξασφαλίσουμε την άριστη ποιότητα της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φαντακανκάμ, λέει πρόεδρος. Εγώ είμαι οικολόγος και προφανώς με ενδιαφέρουν όλα αυτά τα στοιχεία. Μάλιστα. Προθεσμία για την κατάφυση τροπολογίων 12 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με την εκθέση του κυρίου Ισμαήλ Ερτούγκ για την δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς άλλη καθυστέρηση. Σας δίνω το λόγο κύριε Ερτούγκ για να μας προσφέρετε την εκθέση αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πριν από κάποιο χρονικό διάστημα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό για το μέλλον θέμα. Τώρα θα εξετάσουμε τις ε, πρωτοβολίες που υπευλήθησαν. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που μπήκαν στον κόπο να υποβάλουν τροπολογίες. Και έχουμε και τρεις μακροσκελείς ε, νομοδοτήσεις ΙΜΚΟ, ΙΤΡΕ και ΕΝΒΙ. Ξέρουμε ότι Οι μεταφορές είναι υπεύθυνε για ένα μεγάλο ποσοστό των ε, εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και θέλουμε το αργότερο μέχρι το 2005 οι μεταφορές να μην συμβάλλουν καθόλου. Αν εξετάσω αυτές τις τροπολογίες και προσπαθήσω να τις ταξινομήσω σε ομάδες, ασχολούνται με τρία κυρίως θέματα, τα οποία παρουσιάζω. Πρώτον, είναι τα εθνικά ε, σχέδια πλαίσιο. και οι εθνικοί στόχοι. Πρέπει να βρούμε ποια είναι η σχέση μεταξύ της ε, δεσμευτικότητας των στόχων και της ε, επικουρικότητας. Ορισμένοι συνάδελφοι προτείνουν ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει μόνα να καθορίσουν τα, τους στόχους ε, αυτούς και άλλοι θεωρούν ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ρόλο. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει περιθώριο για να ε, καθορίσουν τους στόχους τα κράτη-μέλη, αλλά πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε, ούτως ώστε να είναι αξιόπιστοι και επαληθεύσιμοι αυτοί οι στόχοι. Στο παρελθόν ε, εμπιστευτήκαμε πολύ τα κράτη-μέλη, τους δώσαμε την ευκαιρία αυτοί να καθορίσουν τους στόχους, αλλά ξέρουμε τι συνέβη. Αλλά ε, βεβαίως και η, η προσπάθειά μας πρέπει να επαναπροσανατολιστεί προς μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση τώρα. Όλοι αναφέρονται σε πόσες πιστώσεις πρέπει να υπάρχουν. Η Άλντε θεωρεί, συγγνώμη, όλοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξουν περισσότερες ε, πιστώσεις και ότι όλα αυτά δεν μπορεί να τα επιτύχει μόνο η δημόσια χρηματοδότηση. Πρέπει λοιπόν και οι ιδιωτικοί επενδυτέ και επιχειρήσεις να δεσμευτούν ότι θα συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και τονίζω ότι σε διάφορα κράτη-μέλη υπάρχουν ε, δυνατότητες ε, και έχουμε διαπιστώσει ότι διάφορες επιχειρήσεις σε ένα μικρό επίπεδο ε, χρηματοδοτούν υποδομές Οι περισσότεροι βεβαίω ασχολούνται με ορισμένου τομεί μεταφορών, αλλά κάτι γίνεται. Αυτέ οι προσπάθειε πρέπει να υποστηριχθούν από πλευρά μα ω νομοθέτε. Ποια θα είναι ακριβώ η μορφή τη χρηματοδότηση, έκανα μια, πρόταση. Βεβαίω ε, δεν ξέρω αν συμφωνούν όλοι. Θα πρέπει να το συζητήσουμε, αλλά γενικά υπάρχει ε, γενικά υποστήριξη για τις προτάσεις μου. Τρίτον, επέκταση του τομέα εφαρμογή τη οδηγία. Ε, χαίρομαι γι' αυτό, χαίρομαι που έχω την αναγκαία υποστήριξη. Να περάσουμε και πέρα από την ε, διευκόλυνση ε, συνδέοντα την Ευρώπη στον τομέα των μεταφορών. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα, επέκταση του δικτύου, η δυνατότητα να υπάρχει σωστή φόρτωση, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων, όλα αυτά να είναι επικερδή αλλά και αποδεκτά από τους ε, πολίτες και ο κύκλος ζωής των καυσίμων, όλα αυτά, νομίζω για όλα αυτά δεν έχουμε προβλήματα να βρούμε συμβιβασμούς. Δεν θα έχουμε προβλήματα. Έχω αναφέρει και άλλα θέματα στο παρελθόν και ε, προσλέπω στην περαιτέρω συζήτηση και την έγκριση και σε ευχαριστώ για την εργασία μέχρι τώρα. Ευχαριστώ κύριε Αρτούγκ για την παρουσίαση αυτή ο κύριος Σαλίνη. Θα είμαι πολύ σύντομος. Όπως έχω ξαναπεί σε άλλες επιτροπές όπου ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα, συμμεριζόμαστε τη θέση του εισηγητή, είναι πολύ ισορροπημένη και τα όσα είπε το επιβεβαιώνουν. Έχουμε στη διαθέση μας τώρα πολλές ε, τροπολογίες 131 ε, οι οποίες ε, καταδεικνύουν πόσο ενδιαφέρον είναι το θέμα αυτό για όλο τον κόσμο. Ε, εγώ συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τον εισηγητή, διότι όπως υπενθύμισε ο Ισμαήλ πριν από λίγο, η πρόκληση του θέματος των υποδομών και του θέματος των εναλλακτικών πηγών, των εναλλακτικών συγγνώμη καυσίμων, είναι μια τεράστια πρόκληση ε, και ένα πολύ σημαντικό πολιτικό θέμα. Παρατηρούμε ότι πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δείχνουν να έχουν αποδεχθεί αυτή την πρόκληση επαρκώς. Οπότε το θέμα αυτό το να εξορροπήσουμε έξυπνα ε, τις ευθύνες των επιμέρους χωρών και τα μηνύματα πρέπει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πολλές φορές με τρόπο δεσμευτικό είναι σημαντικό θέμα. Δεν θα είναι κάτι εύκολο εκτιμάμε και εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα μεταξύ όλων των στοιχείων που υπάρχουν ένα στοιχείο το οποίο θα επηρεάσει και τις μεταφορές και τη βιομηχανία. Ε, μας είναι πολύ προσφυλές το θέμα αυτό αφορά την ουδέτερη προσέγγιση που προτείνει και επαναλαμβάνει ο συγγετής σε σχέση με, τις, ε, με τα διάφορα αναλλακτικά καύσιμα. Με τα διαφορετικά αναλλακτικά καύσιμα Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις που προσπαθούν να λαμβάνουν μόνο ένα τέτοιο εναλλακτικό καύσιμο υπόψη. με ένα αντιθέτως μου φαίνεται σημαντικό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πολύπλοκη ε, μεταβατική φάση που θα μας περιμένει. Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε τον δεχόμενο όλων των πιθανών εναλλακτικών καυσίμων και αυτό Μ' αρέσει ε, το ότι επικεντρώνεται σε αυτό η ε, και για τα θέματα των χρηματοδοτήσεων ε, ε, υπάρχουν δύο συναντήσεις οδόν που έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες εβδομάδες, οπότε θα μπορέσουμε να ε, εξετάσουμε τις λεπτομέρειες όλων αυτών των θεμάτων. Γενικά είμαστε ικανοποιημένοι. κύριε Σαλήν ευχαριστούμε. Κύριε με έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και από δικής μου λευρά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή Κατά την ανάγνωση των τροπολογιών διαπίστωσα με μεγάλη μου χαρά και αυτό προκύπτει και από την πρώτη αυτή παρέμβαση στη συζήτηση ότι μοιραζόμαστε και έχουμε ίδιες ανησυχίες με πολλούς συναδέλφους σε ό,τι αφορά τους στόχους για το κλίμα και σε ό,τι αφορά την ε, ανταγωνιστική μας θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν θέλουμε να την εξασφαλίσουμε θα πρέπει ε, γρήγορα να μεταβούμε σε εναλλακτικά τέτοια καύσιμα. Υπάρχουν λοιπόν ε, διάφορα εμπόδια. Τα γνωρίζουμε. Είναι πολύ περιορισμένα τα εναλλακτικά καύσιμα, τα οποία είναι σε σωστή τιμή, σε καλή τιμή και επίσης και οι υποδομές για την ε, προμήθευση, την προμήθεια τέτοιων καυσίμων είναι προβληματική. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια εφαρμόσιμη, ε, λογική και ρεαλιστική λύση ο τομέα των ελεκτικών καυσίμων και των ελεκτικών καυ... οχημάτων στην Ευρώπη είναι νεαρό σε ηλικία. Είναι ακόμα σε εξέλιξη, είναι δυναμικό. Πέρα από τι συγκεκριμένε λοιπόν προτάσεις τις οποίες βρίσκουμε στις ε, τροπολογίε, θα πρέπει βασικά να θέσουμε κάποιες βασικές αρχές ε, για την κοινοτομία, για την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Και άρα θα ήθελα να τονίσω καταρχάς ε, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια δίκαιη και ανοιχτή αγορά για να έχουμε το καλύτερο προϊόν στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχουν πρότυπα, προδιαγραφές και υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την διαλειτουργικότητα μεταξύ των ε, σταθμών ε, προμήθειας καυσίμων και του τελικού χρήστη. Μεσοπρόθεσμα επίσης υπάρχουν διάφορες μεταβατικές λύσεις οι οποίες θα προκύψουν και οι πολιτές θα πρέπει να επιλέξουν το καύσιμο το οποίο τον βολεύει καλύτερα τελικά. Για να μην εξεραστεί λοιπόν καμία τεχνολογία στη διαδικασία αυτή, εμείς ως νομοθέτες θα πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της ουδετερότητας, της τεχνολογικής ουδετερότητας και να τη συμπεριλάβουμε στην έκθεση σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση, συμφωνώ με τον εισηγητή δεν ε, κοιτάμε μόνο τις δημόσιες αρχές, αλλά και τον ιδιωτικό κλάδο. Και ως νομοθέτης νομίζω ότι αυτό που είναι πρώτη τη σημασία είναι να δημιουργήσουμε το σωστό πλαίσιο, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα να επενδύσει και ο ιδιωτικό κλάδο. Και εδώ θα πρέπει να δούμε τι επίπεδο φιλοδοξία θα ακολουθήσουμε, νομική βεβαιότητα και ρεαλισμού φυσικά. Και τέλο, συμφωνώ με κάποιου συναδέλφου ότι κάποια κρατημέλη δεν ανταποκριθήκαν στις υποχρεώσεις του. Και θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να μα περιορίζουν οι στόχοι που έχουμε θέσει. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση μπορεί να αποτελεί, για παράδειγμα, την ε, χορήγηση προτάσεων από, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ τα κράτη-μέλη, λαμβάνοντα υπόψη πάντα φυσικά τι εθνικέ δυνατότητε σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Προσβλέπω στη συνέχιση της επικοδομητικής συνεργασίας μας, γιατί θα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Ο κύριος Ρικέ έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Ισμαήλ. Ήταν εξαιρετική η έκθεση αυτή και εξαιρετικά πολύπλοκη, γιατί είναι πολύπλοκο το θέμα. Δεν ξέρει κανείς από πού να αρχίσει να μελετά αυτό το σύστημα από την αγορά των αυτοκινήτων, από την αγορά ενέργειας. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μάλιστα σε όλους αυτούς τους τομείς μεταξύ των κρατών μελών για λόγους ε, κατά κύριο λόγο που αφορούν ε, την αγορά των αυτοκινήτων παρά την αγορά της ενέργειας. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω και το υπογραμμίζει και ο εισηγητής ότι χρειάζεται τεχνολογική ουδετερότητα, τυποποίηση για τους σταθμούς εφοδιασμού και εναρμόνιση σε ε, ε, ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Αν δούμε το ιστορικό, ε, εμείς φυσικά έχουμε εφεύρει τα αυτοκίνητα με βενζίνη και δίζελ πριν υπάρξουν βενζινάδικα και πρατήρια. Θυμηθείτε τι υπήρχε στις αρχές του 20ου αιώνα. Τα πρατήρια βενζίνης άνοιξαν μετά από την παραγωγή των αυτοκινήτων. Θυμηθείτε τι έγινε στι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη. Εγώ θυμάμαι, λόγω τη ηλικία μου, ότι παλιότερα όταν πηγαίναμε με το αυτοκίνητο στι χώρε τη επωνομαζόμενη Ανατολική Ευρώπη, πριν πέσει ο τείχο, εγώ κυκλοφορούσα με μία κάρτα που είχε, με ένα χάρτη συγγνώμη, που μου ανέφερε πού υπάρχουν πρατήρια που δίνουν βενζίνη σούπερ, διότι ο αριθμό των αυτοκινήτων, η αγορά, οι τύποι των καυσίμων δεν αντιστοιχούσαν σε αυτά που γνωρίζαμε στην Δυτική Ευρώπη. Η αγορά αυτοκινήτων λοιπόν ε, εξαρτάται και από την αγορά πρατηρίων. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι στην εξέλιξη των δικτύων και των αυτοκινήτων ε, θα πρέπει να παρατηρούμε, να προσέχουμε να μην γίνουν κάποια λάθη. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι ότι ο τύπος των αυτοκινήτων θα επηρεάσει ιδιαίτερα τη φύση του δικτύου. σήμερα αν η μέση αυτονομία είναι 160 χιλιόμετρα για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ε, αυτό είναι μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα 400 ή 600 χιλιόμετρα της δεύτερης γενιάς ηλεκτρικών οχημάτων. Όταν υπάρχει λοιπόν επαρκή αυτονομία, εμβέλεια, μπορεί κανείς να πάει πιο μακριά στο δίκτυο. Αλλά τι σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ο ίδιος τρόπος εφοδιασμού. Δεν μιλάω για αλλαγή μπαταριών, ε. δεν νομίζω ότι θα βολέψει κανέναν, αλλά υποχρεούστε να χρησιμοποιήσετε ε, συστήματα ταχείας φόρτισης αν υπάρχει σημαντική αυτονομία, κάτι που απαιτεί ανοικοδόμηση, αναθεώρηση όλου του συστήματος ε, ανεφοδιασμού. Σε αυτό έχω επιμείνει και εγώ στις τροπολογίες μου. Θα πρέπει να αφορούν πολλαπλές μορφές ενέργειας ε, τα πρατήρια. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλο σταθμό για το υδρογόνο, άλλο για το αέριο, άλλο για το ηλεκτρικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πιστεύω. Είναι πιθανότατα αυτή η μόνη οδός ε, για το μέλλον, διότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς προς τα πού θα κινηθεί η αγορά ο χρόνο απόσβεση ενό αυτοκινήτου και μια τεχνολογία είναι χρόνια, αλλά ο χρόνο απόσβεση ε, δικτύων είναι δεκαετίες. Οπότε εκεί έχουμε πολλά προβλήματα. Και το τελευταίο που ήθελα να τονίσω είναι ότι η απόψη επενδυτική, μιλάμε για δημόσιε επενδύσει. Εγώ δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν είναι θέση των κρατών να διαθέσουν χρήματα για την ανάπτυξη αυτών των δικτύων. Είναι δίκτυα ιδιωτική πρωτοβουλία. Μπορούμε να βοηθήσουμε και εκεί πιστεύω ότι το FC2 ή το Invest Europe, αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το θέμα παρά το Connecting Europe, το οποίο δεν είναι κατάλληλο ούτε σε οικονομικό ούτε χρηματοοικονομικό ε, επίπεδο. Σίγουρα θα υπάρξει και κάποια κερδοφορία στα δίκτυα, αυτή, στα δίκτυα αυτά. Οπότε αυτοί που θα τα δημιουργήσουν πρώτοι θα κερδίσουν τα περισσότερα, αλλά μέχρι εκεί θα υπάρξουν κάποιε δυσκολίε. Η αγορά λοιπόν των αυτοκινήτων θα καθορίσει την αγορά του ανεφοδιασμού. Είναι κάτι πιστεύω το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε να υπογραμμίζουμε και να μην πιστεύουμε ότι η αγορά των αυτοκινήτων ε, σταματά, ανακόπτεται λόγω της απουσίας ε, πρατηρίων ε, και δικτύων. Κατά τα άλλα, η έκθεση πιστεύω είναι εξαιρετική. Εξαιρετική αφορά έναν ορίζοντα πολύ περίπλοκα, ένα σε πολύ περίπλοκο θεμάτων ε, οικονομικών και τεχνολογικών και σίγουρα δεν θα πρέπει να πάψουμε να προσανατολιζόμαστε προς αυτά τα αυτοκύματα. Το λόγο έχει ο κύριος Keith Taylor. Ευχαριστούμε κύριε Ρικέ. Ο κύριος Keith Taylor, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που ε, είμαστε πάλι εδώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ερτούγ. Θαυμάσια εκθεσίως τώρα. Περιμένουμε βέβαια ακόμη τις συμβαστικές, αλλά εγώ προσβλέπω στη συνεργασία με άλλα μέλη για να υπάρξει συμφωνία στις ε, επικείμενες ε, συζητήσεις των σκιωδών. Θα παρουσιάσω κάποιες από τις τροπολογίες μας και θα θέσω ορισμένα θέματα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για μας ε, θέμα κλειδί είναι ο κύκλος ζωής των εκπομπών να ε, λαμβάνει υπόψη σε οποιαδήποτε αποτίμηση των εναλλακτικών καυσίμων. Για να λύσουμε το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής πρέπει να αποφύγουμε, να επιδεινώσουμε κάποια προβλήματα μέσω κάποιων πολιτικών για εναλλακτικά καύσιμα. Για παράδειγμα, κάποιες, ε, κάποια, εναλλακτικά, κάποια λεγόμενα εναλλακτικά καύσιμα είναι ορυκτής προέλευσης. Για παράδειγμα, μέσω του σχιστολιθικού ε, αερίου ή του ε, ε, φινικελαίου. Όλα αυτά μπορεί να έχουν σοβαρά προβλήματα για την ίδρυυση, για τη χρήση της γης, για το περιβάλλον και φυσικά και για τους πολίτες. <clears throat> Άρα, ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει κριτήρια βιωσιμότητας, ούτως ώστε να εκτιμήσουμε σωστά και να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις. Επίσης πρέπει να υπάρχει βιώσιμη πολιοδομία. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το θέμα αυτό στις επικείμενες συζητήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επιπλέον 800 εκατομμύρια. Κυρίως πρέπει να εστιαστεί αυτή η χρηματοδότηση στη στήριξη της υποδομής των εναλλακτικών ε, καυσίμων για τις δημόσιες μεταφορές, ούτω ώστε να αυξηθεί η κινητικότητα μέσω λεωφορείων, τραμ, τρένων και ε, ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων. Για τη χρηματοδότηση, όπως και ο κ. Ρικέ, δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν ε, τροπολογίες που να καλούν για επιπλέον δημόσιες χρηματοδοτήσεις για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων. Και ελπίζουμε να ληφθούν υπόψη και οι διαφορές ε, της φορολόγησης των διαφόρων ε, μορφών μεταφορών. Αυτό πρέπει να το εξετάσουν τα κράτη-μέλη και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, πόσο ρεαλιστικές θεωρείτε ότι είναι οι υποσχέσεις του κυρίου Γιούνκερ προς τον κύριο Τραμπ να ε, εισαχθούν ε, τεράστιες επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου. Και αυτό το εισαγόμενο αέριο θα δημιουργηθεί από υδρορογμάτωση στις ΗΠΑ και θα χρειαστούμε και επιπλέον τερματικά αερίου και αν ναι ποιος θα τα πληρώσει και πώς θα γίνει κατόπιν η διανομή αυτού του αερίου. Βεβαίως θα συνεργαστώ με τους άλλους ε, σκιώδεις για να καταλήξουμε σε μια τελική έκθεση που θα βοηθήσει πραγματικά τα κράτη-μέλη ούτως ώστε ταχαίως να <clears throat> αποφευχθούν να ε, έχουμε δημόσιες μεταφορές που να μην παράγουν οξυδία του άνθρακα. Και προσβλέπω στις πρώτες συζητήσεις που πιστεύω θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τέιλορ. Τώρα πρέπει να δώσω περιορισμένο χρόνο γιατί κατόπιν έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Ήτρε και ήδη έχουμε καθυστερήσει. Γοβονταλόν, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Ερτούγκ και τους Κιώδης για τις παρεμβάσεις τους το θέμα αυτό είναι ευρωπαϊκό. Τα αυτοκίνητα δεν σταματάνε στα σύνορα και ούτε και το διοξείδιο του άνθρακα. Είναι θεμελιώδες θέμα για την κινητικότητα του αύριο. Αλλά όπως ήδη υπόθηκε, το χρονοδιάγραμμα δεν είναι το βέλτιστο, γιατί προχωράμε προς το τέλος της θητείας και έχουμε μόνο μια έκθεση πρωτοβουλίας. Θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο προχωρημένοι, να υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία κατάλληλη. Έχει να κάνει και με τη βιομηχανική μας βάση το θέμα αυτό, αλλά όπως είπε και ο κύριος Κριστέλιο, έχει να κάνει και με τις διεθνείς γεωπολιτικές ισορροπίες, έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, που θέλουν να είναι σίγουροι ότι θα μπορούν να φορτίζουν τα οχήματά τους όπου και αν πάνε. Και έχει να κάνει επίσης και με την καινοτομία και με ε, διάφορες γεωργικές παραγωγές. Όλα αυτά τα θέματα δεν μπορούμε να τα ξεπετάξουμε το δίκτυο ε, διανομής των ε, εναλλακτικών καυσίμων δεν επαρκεί τώρα, αλλά τι θα πρέπει να γίνει και μέχρι πότε, όλα αυτά είναι υποσυζήτηση. Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, μάλλον να τεθεί, να ξεκινήσει. Και οι ε, δυνατόν πριν ξεπεράσουμε τους δύο βαθμούς Κελσίου θέρμανση του πλανήτη. Πρέπει να έχουμε τα αναγκαία μέτρα για να σεβαστούμε τις συμφωνίες των Παρισίων και να έχουμε και πρωτοπόρα θέση. Πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση και μια στρατηγική που να διασφαλίσει τη συνένεση. Πρέπει το θέμα αυτό να αποτελέσει απόλυτη προτεραιότητά μας και όχι βεβιασμένα μαζί με όλα τα άλλα θέματα που εκκρεμούν στον τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ κυρία Γονταλόν. Ο κύριος Πέτερ Λούγκρεν. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, τα εναλλακτικά καύσιμα είναι θέμα μέλλοντος. Ήδη υπάρχουν, πρέπει να υπάρξουν περισσότερα. Ακόμη και για τα αγωνιστικά μου ε, αυτοκίνητα χρησιμοποιώ διάφορα αλκαλικά. Ως μέλλον της Επιτροπής Μεταφορών προσπάθησα να αγοράσω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το αγόρασα, έχει 30 κιλοβάτ μπαταρία και λειτουργεί μια χαρά ιδιαίτερα στην Ήπεθρο. Μπορεί κανείς να το βάλει στην πρίζα και να το φορτίσει. Ενώ στην πόλη ε, δεν είναι εύκολο να τα φορτίσουμε. Είναι δυνατόν να έχω τόσο μακριά μπαλαντέζα που να το βάλω σε μια πρίζα στο σπίτι μου και να κρέμεται από το μπαλκόνι. Αλλά στην Ήπεθρο είναι πιο εύκολο. Νομίζω ότι είμαι ο μόνος στην Επιτροπή Μεταφορών που οδηγώ ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Βεβαίως, ε, στην Ήπεθρο λειτουργούν όλα αυτά. Ο κύριος Φαν Μίντεμπουργκ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σα ευχαριστώ. Ελπίζω να μου δώσετε και λίγο χρόνο παραπάνω, γιατί μιλάω και εξ ονόματο τη κυρία Γκιζίν Μέισνερ, η οποία είναι σκιώδη στο θέμα αυτό. Δεν μπόρεσε όμω να παραβρεθεί. Η Γκιζίν, λοιπόν, υποστηρίζει του φιλόδοξου στόχου για το LNG ε, σε προηγούμενη θητεία, όταν ε, έγινε η διαπραγμάτευση τη οδηγία για τα εναλλακτικά καύσιμα. Το LNG εξακολουθεί φυσικά ε, να αποτελεί ρηκτό καύσιμο αλλά όσο δεν υπάρχουν πλήρη εναλλακτικές, πλήρες εναλλακτικές, θα πρέπει να υποστηρίξουμε και το LNG. Το ευρωποιημένο αέριο. Επίσης, σε ό,τι αφορά και τα πλοία που χρησιμοποιούν LNG, υγροποιημένο αέριο, θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια και σε παγκόσμιο επίπεδο οι στόχοι θα είναι από 3,5% σε 0,5%. Άρα θα χρειαστούμε ακόμα πιο πολλά πλοία ε, που θα χρησιμοποιηθούν, ε, που θα χρησιμοποιούν ε, υγροποιημένο αέριο, όχι μόνο στη Βαλτική και στη Βόρεια Θάλασσα. Ένα άλλο θέμα, οι φόροι για την ενέργεια, ιδιαίτερα για τον ηλεκτρισμό. Είναι πιο φτηνό να παράγεται ηλεκτρισμός με τους κινητήρες των πλοίων πάνω στο πλοίο παρά να συνδέονται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Και άρα ένα μεγάλο τμήμα της ηλεκτρισμού δεν χρησιμοποιείται και αυτό προφανώς δεν βοηθά ε, σε ό,τι αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση στους ευρωπαϊκούς λιμένες και σε ό,τι αφορά το θέμα τη έλλειψη της εφαρμογής ε, της οδηγίας Είναι θέμα αυτό, θεωρεί η Γκυζίνα, γιατί κοιτώντα ποιες πόλεις και ποιες χώρες έχουν εφαρμόσει και έχουν υλοποιήσει τους στόχους της οδηγίας, τα πράγματα είναι προβληματικά. Άρα αυτό θα υποστηρίξει η Γκυζίνα. Δέκα δεύτερα για προσωπικές ε, παρατηρήσεις. Κύριε Έρτουγκ, και εγώ υπέβαλα κάποιες τροπολογίες θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ε, επιλέξουμε τη λύση μια, ενός νέου ταμείου, να μην κάνουμε μικροδιαχείριση. Θα πρέπει να αποφύγουμε προνομιακή θέση. Δεν με ακούτε, άρα ούτε εγώ είμαι σε προνομιακή θέση. Κύριε του λέω. Ελπίζω να σημειώνετε αυτά που λέω. Γιατί νομίζω ότι καλά θα κάνετε να μην ακολουθήσετε αυτά που λέτε στην παράγραφο 7. Να μην γίνεται δηλαδή μικροδιαχείριση, να δημιουργηθεί ένα νέο ταμείο και κατά τρίτον. Να υπάρχουν κάποιοι φορείς οι οποίοι θα έχουν προνομιακή μεταχείριση χωρίς να είναι σαφές όμως πόσο θα πρέπει να συνεισφέρουν στο ταμείο αυτοί οι παράγοντες. Άρα κοιτάξτε το λίγο το θέμα αυτό, γιατί αυτό αποτελεί πρόβλημα όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για τμήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φαμίλτεμπερ, λέει Πρόεδρο. Ο κύριο Βερντούνι, πού είναι? Η ε, κυρία Κλερτεπρέ, έχει το λόγο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Έχετε το λόγο λοιπόν για δύο λεπτά για να μας απαντήσετε. Πολύ γρήγορα λοιπόν να σας πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε αυτό το θέμα και από τις πολυαριθμές τροπολογίες ε, φαίνεται πόσο ενδιαφέρει το θέμα την Επιτροπή. Υγούμαστε λοιπόν του μέλλοντο τη κινητικότητα στην Ευρώπη. Δύο παρατηρήσει από πλευρά μα. Έχουμε συζητήσει αυτή την ισορροπία μεταξύ εθνικού επίπεδου και ευρωπαϊκής παρέμβαση. Έχω αναφέρει επανειλημμένω ότι σύντομα θα αρχίσουμε να αξιολογούμε πιο συστηματικά την οδηγία. Δεν θα αξιολογούμε μόνο το εθνικό πλαίσιο πολιτική, αλλά και την ίδια την οδηγία βασισμένη σε αυτή την προτιάσκηση των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι θα προσπαθήσουμε επίσης να εξετάσουμε τα διάφορα εναλλακτικά καύσιμα και πώς σχετίζονται με συγκεκριμένους τρόπους μεταφορών. Από αυτή την άποψη θα ήθελα να ε, επαρέλθω σε αυτό που είπε ο κύριος Βαν Ο κύριος Ρικέ ανέφερε αυτό το ζήτημα του κότας και του αυγού, ποιος είναι ο οδηγός ουσιαστικά, ποιος ηγείται της μετάβασης προς την ε, κινητικότητα μηδενικών εκπομπών. Έχετε δίκιο που το λέτε και το αυτοκίνητο έχει να παίξει σημαντικό ρόλο. Μέχρι να υπάρξει επαρκής προσφορά και προς τον καταναλωτή, όσο δίκτυο και να φτιάξουμε πρατηρίων δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Αληθεύει όμως επίσης ότι για να γίνει αποδεκτή τεχνολογία από τους καταναλωτές θα πρέπει να είναι και αυτοί βέβαιοι ότι υπάρχει το δίκτυο. Οπότε έτσι θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε ολόκληρο το οικοσύστημα. Η μεταφορά της οδηγίας, να σας πω μια καλή είδηση. Είχαμε αναφέρει ότι παρακολουθούσαμε προσεκτικά τη μεταφορά της οδηγίας. Όλο και περισσότερα τώρα κράτη-μέλη έχουν υπακούσει, για να το πω έτσι, τους κανόνες και έχουν ε, ε, προβεί σε εφαρμογή στην παρουσιαφάση. Τι άλλο ήθελα να πω, να δούμε λίγο το ποιος θα πληρώσει τις υποδομές. Και αυτό που ήθελα να πω εδώ ήταν ότι πρώτα ε, στις πρώτες του μέρες η διευκολύνση συνδεδεμένες στην Ευρώπη ε, έλαβε συμβολή από εμάς. Ε, μέσω, ε, συγγνώμη, δώσαμε εμείς συμβολή για τις υποδομές μέσω χρηματοδοτήσεων, αλλά μετά η αγορά σταδιακά και έτσι χρησιμοποίησαμε το συνδέοντα την Ευρώπη και με καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και αυτό ήθελα να τονίσω ότι όλο και περισσότερα έργα τώρα έχουν φτάσει σε σημείο ορίμαση τέτοιου που μπορούν εκεί να χρησιμοποιηθούν τα καινοτόμα μέσα και το μελλοντικό εμβέστηγιο. Το τελευταίο που θέλω να αναφέρω, πολλές τροπολογίες που υπάρχουν εδώ, αμφισβητούν κάπου το επίπεδο φιλοδοξίας στον τομέα. Και αυτό που θέλω να πω και το αναφέρετε και πολύ. είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης σε αυτό τον τομέα. Πρέπει να κινηθούμε στον τομέα αυτό και να προοδεύσουμε και σε θέματα δεξιοτήτων. Σίγουρα ο τομέας αυτός χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις από εμάς και από τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις θέσεις εργασίας. Ευχαριστή Πρόεδρος. Ευχαριστούμε Κλέντε Πρέ από την Επιτροπή. Τον τελευταίο λόγο έχει ο κύριος Ερτούγκ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε ούτε μία από τις τρεις ερωτήσεις που της έθεσα. Και θα ήθελα, παρακαλώ, Πρόεδρε, να με βοηθήσετε, γιατί θα ήθελα να πάρω κάποιες απαντήσεις, λέει ο κύριος Τέιλορ. Είχα δώσει τέσσερα λεπτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν μας απάντησα. Αλλά τώρα και εμείς έχουμε καθυστερήσει για την επόμενη συζήτηση. Άρα το λόγο έχει ο εισηγητής μας. Και η κυρία Κλέρτε Πρέ, παρακαλώ να απαντήσει στον κύριο Keith Taylor. Αν δεν λάβει απαντήσει ο κύριο Τέιλορ, θα φροντίσουμε εμεί να ζητήσουμε να μα απαντήσει. Γραπτά η κυρία Ντεπρέ. Κύριε Ερτούκ, θέλετε το λόγο για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή συζήτηση για την έκθεσή σα. Και μετά να πω και τι προθεσμίε για την κρατήση τροπολογιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου, λέει ο κύριο Ερτούκ, για τη συμμετοχή του και αποδεικνύεται εκ νέου ότι θα καταφέρουμε να βρούμε εκείνο τόπο. Παραδέχτηκα του σε θέματα χρηματοδότηση το θέμα που με απασχολεί δεν είναι να επανεφεύρουμε τον τροχό ή να δημιουργήσουμε απαραίτητα κάτι καινούριο ίσα ίσα για να πούμε ότι κοιτάξτε τι φτιάξαμε. Όχι, το θέμα είναι το εξή. Όταν ψάχνουμε μία λύση, έναν δρόμο, ένα μηχανισμό για την ανάπτυξη τέτοιων υποδομών, να υποστηρίξουμε την όλη διαδικασία. Και με χρηματοδότηση προφανώς. Εδώ να πω ότι την τελευταία περίοδο ως ε, εισηγητής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τότε συμπεριέλαβα τη διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη και κάθισα και κατάλαβα ότι τότε με την ε, οργάνωση, με την υπηρεσία η νέα έχουμε μάλλον στο πρόσωπο της εταιρείας αυτής, της υπηρεσίας αυτής, έναν αρμόδιο παράγοντα για την δημιουργία σχετικής πλατφόρμας, ε, για την, ε, τον καθορισμό Ευρωπαίων συντονιστών. Έχουμε δυνατότητες λοιπόν. Είναι λοιπόν ε, ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι κινούνται τα ευρωπαϊκά Θα πρέπει να επενέσουμε εκείνους οι οποίοι βάζουν το χέρι στην τσέπη σε εποχές που τα πράγματα είναι ακόμα επικίνδυνα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις αυτές. Είμαι και πολύ ανοιχτό σε οτιδήποτε μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον. Είναι προφανώς καινούριο και το θέμα, το θέμα αυτό και περιμένουμε πολλά να γίνουν ακόμα και στο μέλλον, αλλά ως τώρα ε, είναι πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 24 ε, Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας και να καλέσω τους... Ε, μάλλον να, προσ... να καλωσορίσω τους συναδέλφους από την Επιτροπή Ήτρε και τα λέμε σε 5 λεπτά. Κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για 5 λεπτά.